καλωσορίζω, και σά και σας και τους εμπειρογνώμονες μας πρώτα και καλύτερο τον κύριο Ματσόνε. Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης της Ευρωβίζιας και τον πρώην συνάδελφό μας Νατσουγκάιντε Γκάντενς που ήταν μέλος και της Επιτροπής μας και τώρα είναι πολύ σημαντικός παράγων στο EBU. Είναι και ο κύριος Κλόντερικ Πορού από την οργάνωση Europe Cinema και ο Αντώνιος Σουάρες, Γενικός Γραμματέας της Αιγίδας. Καλωσοριστείτε όλοι. Να σας πω πώς οργανώνουμε την ακρόαση. Ένας γύρος παρουσιάσεων, κάθε εμπειρογνώμων θα μιλήσει 10 ολόκληρα λεπτά. Και μετά ερωταπαντήσεις 45 λεπτά, συζήτηση δηλαδή με άλλα λόγια. Μετά εμπειρογνώμονες άλλα 5 λεπτά ο καθένας για να απαντήσουν. Και τέλος θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν και στην Πολωνική Προεδρία που παρίστανται αμφότερες. Θα σας υπενθυμίζω τα τεχνικά θέματα. Οι συνεδριάσεις αναμεταδίδονται ηλεκτρονικώς. Όλοι μπορούν να σας δουν, σας παρατηρούν, σας παρακολουθούν. Να φέρεστε όπως πρέπει. Η κάμερα συνήθως ε, κάνει zoom στον ομιλητή. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί μικρόφωνο αριστερά του. Αριστερά του. Τα λέω αγγλικά γιατί αγγλικά τα ετοίμασα, αλλά η μητρική μου γλώσσα είναι τα γερμανικά. Γερμανικά. Το θέμα της ψηφιοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία και διατήρηση του Ευρωπαϊ... της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Διαθέτει το περιεχόμενο δηλαδή online. Γι' αυτό οργανώσαμε αυτή την ακρόαση σήμερα. Ως Ευρωπαίοι αλλά και ως ενωσιακοί Θέλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να τονιστεί πολύ περισσότερο ο πολιτισμός στην όλη συζήτηση περί Ευρώπης. Μιλάμε πάντοτε για λεφτά, για κρίσεις, αλλά συνήθως ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός είναι η βάση της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης και θα έπρεπε να ληφθεί αυτό σοβαρά υπόψη. 96 δισεκατομμύρια και πάνω από χίλια ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο. Πολλές αλλαγές έχουν σημειωθεί στον τομέα αυτόν την τελευταία δεκαετία. Η ψηφιακή τεχνολογία ήδη κατέστησε πιο πρόσβατα τα ευρωπαϊκά έργα και εκτός Ευρώπης και δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες όπως το Video On Demand. Είναι όμως ακόμη ασαφής η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται αυτές οι εξελίξεις. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από κατακαιρματισμό και πολιτιστικό και βιομηχανικό και γι' αυτό βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή και ζητήσαμε από το συνάδελφό μας Μπόρις να μας γράψει μια έκθεση για αυτό το θέμα και για να υποβοηθηθεί προβλέψαμε και αυτή την ακρόαση. Έχουμε πολλές προκλήσεις και νομικές και πολιτιστικές και πολλές από αυτές είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Το ίντερνετ και η ψηφιακή διάδοση περιεχομένων δημιούργησαν νέες προκλήσεις στον οπτικοακουστικό τομέα αλλά και νέες δυνατότητες και ευκαιρίε. Πολλές φορές οι ηθοποιοί και οι άλλοι παράγοντες του πολιτιστικού τομέα αντιτίθενται στις αλλαγές αυτές αλλά υπάρχουν και οι προτάσεις της Κομισιόν πρόσφατα για την αντιμετώπιση της δυσκολίας του θέματος των δικαιωμάτων. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη δημιουργία ε, μιας πραγματικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς οπτικοακουστικού περιεχομένου για να προωθηθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία. Και γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν νέες αγορές ώστε η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας να διαχέεται παντού ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν όπως πρέπει την ψηφιακή εποχή και προσβλέπουμε με μεγάλη ανυπομονησία σε αυτά που θα μας πούν οι εμπειρογνώμονες γιατί είμαι σίγουροι ότι θα ακούσουμε πολλά χρήσιμα πράγματα. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Τζάκομο Ματσόνε, Γενικό Γραμματέα της Ευρωβιζιόνε. Ορίστε, έχετε το λόγο κύριε Ματσόνε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ. Και επειδή είμαι Ιταλός θα μιλήσω στη γλώσσα αυτήν. Παρακαλώ κρατήστε τα ακουστικά σας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Ε, ε, για λόγους ε, πολιτιστικής διαφοροποίησης και επικοινομορφής θα μιλήσω στα Ιταλικά. Η πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα, ένα από τα βασικά ε, αντικείμενα της δουλειάς μου. Ασχολούμαι εδώ και 25 χρόνια με το θέμα αυτό, ε, ξεκινώντας τη ΡΑΗ, τότε πρώτο ξεκινήσαμε τα Euronews ε, και τώρα απασχολούμαι, όπως ακούσατε, στην, στην EBU. Υπάρχει λοιπόν όλη, αυτό, το, όλη αυτή η βεντάλια απασχολήσεών μου και νομίζω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο οι δημόσιοι φορείς στην Ευρώπη. Είναι ένας καθοριστικός ρόλος ε, που ήταν ίσχυε στο παρελθόν αλλά θα ισχύσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον που θα είναι ψηφιακό. Ε, θα ήθελα να ε, παρουσιάσω λιγάκι το πρόβλημα. Πράγματι, πέρυσι, εκ μέρου ε, τη δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη, είχαμε 10 εκατομμύρια επενδύσει σε πρωτότυπα προγράμματα και αυτό το ποσό δεν έχει αλλάξει, παρότι πέρυσι ήταν μια χρονιά με πάρα πολλέ οικονομικέ δυσκολίε για πολλά μέλη μα. Η τηλεόραση, ακόμα και σήμερα, είναι ένα μέσο επικοινωνίας πολύ δυνατό ο χρόνος ε, τηλεθέασης ε, έχει αυξηθεί πάνω από 3,5 ώρες την ημέρα ανάτομο. Και η καινοτομία είναι ότι υπάρχει νέο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο πλέον προσφέρεται online. Όχι όπως ε, είχε προβλεφθεί στην οδηγία που εγκριθήκε πριν από δύο χρόνια. Το 2010 είχαμε 5 δις υλικό ε, βίντεο που κατέβηκε στη Μεγάλη Βρετανία και σε μεγάλο βαθμό ήταν υλικό το οποίο είχε ε, παραχθεί από τον τομέα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι χρόνοι τηλεθέασης αυξάνονται ε, και αυτό αφορά μόνο το τι βλέπει κανείς στην τηλεόραση. Όταν μιλάμε για τη συνεισφορά των ε, δημόσιων υπηρεσιών στην ε, παραγωγή και στο πρωτότυπο περιεχόμενο, βλέπετε ότι ένας από τους ε, βασικούς στόχους της οδηγίας τηλεόραση χωρίς σύνορα ήταν να διασφαλιστεί ευρωπαϊκή παραγωγή που θα, που εκπέμπεται και από την τηλεόραση. Αυτό το γράφημα είναι, λέει πάρα πολλά από μόνο του. Το 2009 βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι που αφορά την ίδια παραγωγή ή την ανάθεση παραγωγής σε ανεξάρτητους παραγωγούς. Αριστερά στο διάγραμμα βλέπετε το BBC το οποίο εκπέμπει, έχει πολλές παραγωγές και βλέπουμε ότι ε, σιγά σιγά μειώνει το ποσοστό ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Ε, μπορούμε στο γράφημα να δούμε τις ε, δαπάνες και τους πόρους ε, και όσο περισσότερο είναι η πόρη τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ποσοστά παραγωγής. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε η ψηφιακή ατζέντα στην Ευρώπη εμείς ως broadcasters, ως άτομα του τομέα δείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πιστεύουμε ότι η ψηφιακή πρόκληση είναι πλέον η ευκαιρία για να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν βαίνουν καλώς αυτή τη στιγμή και κυρίως για να ληφθεί υπόψη ε, ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες ε, οι οποίοι εντάσσονται σε έναν ενιαίο χώρο και μερικοί είναι μεγάλοι, άλλοι μικρότεροι, μερικοί με περισσότερους πόρους, άλλοι με λιγότερους. Αυτό είναι το βασικό γράφημα που δείχνουμε για να παρουσιάσουμε την ε, ψηφιακή ατζέντα. Αν ψάξετε τη λέξη προγράμματα δεν θα τη βρείτε. Θα βρείτε μια λέξη που λέει περιεχόμενο. Ε, περιεχόμενο είναι ουδέτερη η λέξη αυτή γιατί προγράμματα είναι αυτές οι ειδήσει που βλέπουμε κάθε μέρα ε, το πρόγραμμα Μεγάλος Αδελφός ε, είτε μας αρέσει όχι όλα αυτά που έχουν σχέση με την πολιτική στις χώρες μας εδώ όμως βλέπουμε ότι όλα αυτά περιορίζονται σε περιεχόμενο σαν να πρόκειται για την βενζίνη που χρειάζεται για να κινηθεί ένας κινητήρας δυστυχώς η στάση ε, της ε, παραγωγικής, του παραγωγικού τομέα είναι στάση ουδέτερη ε, και λέει ότι για να λειτουργήσει το όλο θέμα πρέπει να υπάρχει και η τροφοδοσία. Εγώ είμαι πεπισμένος ε, και αυτό ισχύει και για όλους του φορεί του οποίους δούλεψα, ισχύει το αντίθετο. Αυτό το γράφημα είναι λάθο. Εμεί πρέπει να παράγουμε ποιοτικά προγράμματα στην υπηρεσία των πολιτών, στην υπηρεσία της κοινωνική συνοχή. συνοχής. Δεν μπορούμε να παράγουμε προγράμματα απλά και μόνο για να λειτουργεί ένα ε, φαύλο κύκλο. Ε, σύγκληση. Δυστυχώς η στάση που επικρατεί όμω είναι διαφορετική. Εδώ λοιπόν η Επιτροπή Πολιτισμού έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Όλη η δουλειά που κάνατε τα τελευταία χρόνια, η έκθεση Μπελέκ με την οποία εργαστήκαμε πάρα πολύ, η έκθεση για τις ε, δημιουργικές, και τους δημιουργικούς τομείς, ε, η έκθεση για την συμβολή των πολιτών το περιεχόμενο των προγραμμάτων, η έκθεση Μπόρις που πρόκειται να παρουσιαστεί. Όλα αυτά έχουν ως στόχο να αλλάξει αυτή η στάση, να είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορούμε ε, να αντιμετωπίζουμε τα προγράμματα κάτω από αυτή την προοπτική που είναι πολύ απαξιωτική. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Το πρόβλημα είναι ότι ο δικός μας τομέας δεν είναι αποκλειστικά τομέας που έχει αφαιθεί στην αγορά. Για πάρα πολλούς λόγους είναι ένας τομέας καθοριστικής σημασίας γιατί συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατία, με τη σχέση με τον ε, πολίτη, η σχέση του πολίτη με τους θεσμούς και έχει ο τομέας αυτός άμεση σχέση και με πολλά άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα δηλαδή πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά παραγόντων οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν την εξέλιξη στο σύνολό της χωρίς να ε, λησμονούνται τα, οι βασικοί στόχοι που είναι η εκπαίδευση του πολίτη και πάρα πολλά άλλα συναφή. Έτσι λοιπόν ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή ε, Πολιτισμού ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Επιτροπής Πολιτισμού γιατί η Επιτροπή Βιομηχανίας ασχολείται με άλλα πράγματα που είναι εκτός δικτύων. Εσείς όμως ασχολείστε με τα ίδια τα δίκτυα. Κατόπιν τούτου, τα επόμενα χρόνια, οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να υπάρξει πλήρη σύγκληση των προγραμμάτων και πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι καθοριστική σημασία. Παραδείγματος χάρη το δίκτυο ουδετερότητα, neutrality. Ε, η συζήτηση ε, κατ' ουσίαν ε, θα πρέπει να αφορά ένα βασικό θέμα. Σήμερα έχουμε κανάλια ε, τα οποία είναι εξειδικευμένα. Οι πολίτες έχουν συνηθίσει να πατάνε ένα κουμπί και να έχουν αμέσως μια υπηρεσία. Τώρα, όσον αφορά το διαδίκτυο που ε, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, ε, στο διαδίκτυο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει κανείς να κάνει την πλοήγηση για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα δηλαδή τα προγράμματα θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα, προσιτά, εύκολα ε, να μην υπάρχει κανός είδους μπλοκ και να μην ξεχνάει κανείς ένα βασικό στοιχείο που είναι το στοιχείο της δημόσιας υπηρεσίας και το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα. Όχι μόνο λίγοι, όχι μόνο εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα, ε, ειδικέ ε, δυνατότητες ε, να πληρώνουν την τηλεόραση με συνδρομή. Όχι, τα προγράμματα πρέπει να είναι ανοιχτά για όλους τους πολίτες. Ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα, σημαντικό αυτό γιατί θα έχετε πέντε δυνατότητες δυνατότητες να επανέλθετε στο θέμα αυτό. Ένα άλλο λοιπόν σημαντικό επιχείρημα είναι το ε, copyright. Αυτό έχει άμεση σχέση και με τα ορφανά έργα. Ε, εγώ άκουσα τη λέξη προηγουμένω και εντράτω με τις πληροφορίες για να τα επαναλάβω. Όσον αφορά το copyright υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Το copyright ε, είχε προκύψει ως ιδέα σε άλλες εποχές ε, και χαρακτηρίζεται από ένα γραμμικό κόσμο. Όταν όμως ε, η κατάσταση δεν είναι πλέον γραμμική και η σύγκληση είναι ο κανόνας, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή και στο copyright. Πρέπει να υπάρχουν συλλογικέ άδειε, ή δυνατότητα ε, του ψηφιακού διαβατηρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μετάδοση και για να αντιμετωπιστεί και η πειρατεία. Ε, νομίζω ότι εξάντλησα το χώρο που μου είχατε διαθέσει, αλλά βεβαίως αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Και το μόνο που θέλω να πω είναι η υβριδιακή τηλεόραση, hybrid television. Αυτή θα είναι πραγματικότητα από εφέτος, ε, θα διανέμεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και έτσι λοιπόν δημιουργεί αυτή ένα πρόβλημα σε εμά και στο νομοθέτη για το ποιο σύστημα θα κυριαρχήσει και θα εφαρμόζεται. Σήμερα ως έχουν τα πράγματα υπάρχουν οι κανόνες ε, που ισχύουν ε, για την οθόνη και ένα άλλο σύστημα που ισχύουν ισχύει για αυτά που εκπέμπει το διαδίκτυο. Άρα δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς ε, βεβαίως ε, θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύουν οι κανόνες της ε, τηλεόρασης γιατί είναι πιο ασφαλής για τον πολίτη. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ και το συγγνώμη που υπερεύει το χρόνο μου. Ευχαριστούμε κύριε Ματσόνε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον, στην Αντιπρόεδρο της Νόκια στον κύριο Έκη Ορμάλα. Παρακαλώ, στον κύριο Έκη Ορμάλα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω στην σημαντική αυτή εκδήλωση σήμερα. Θα αρχίσω με ένα ευρύτερο θέμα. Στις ε, ψηφιακές βιομηχανίες έχουμε κάποιες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενε τέτοιε βιομηχανίε. Δεν υπάρχει άλλο που έχει τέτοια διψήφια ανάπτυξη σε, σε, στα δεδομένα χρόνια, έτσι όπω ε, ε, έχουν οι συνθήκε, όπω έχουν οι τιμέ και έτσι παράγουμε, δημιουργούμε θέσει εργασία και επομένω ε, είναι ένα ατού που έχουμε στα χέρια μα, ώστε να συνεχίσει η Ευρώπη να έχει αυτήν την ευημερία και κοινωνική συνοχή. Επομένω, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά υποφέρουμε στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε ενιαία αγορά για τις ψηφιακές υπηρεσίες και έχουμε πασχίσει με εμπειρικούς τρόπους να καταλάβουμε το κόστος του να μην υπάρχει ενιαία αγορά για ψηφιακές υπηρεσίες και καταλήξαμε στα στοιχεία τα οποία υπήρχαν τέλος δεκαετίας του 80 που έγινε η αγορά. Επομένω θα μπορέσουμε να πετύχουμε επιπλέον έσοδα 500 δις ευρώ. Εάν μέχρι το 2015 έχουμε ενιαία αγορά θα μπορούσαμε να βγούμε από τη σημερινή κρίση με τα επιπλέον αυτά έσοδα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αυτά τα θέματα δεν βρίσκονται στην κορυφαία προτεραιότητα σε αυτού που πάνε τι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα μπορούσαμε να βρούμε όλα αυτά τα χρήματα και θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει τη χρηματοοικονομική κρίση χωρίς ενή αγορά. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και επομένως θα πρέπει να μπορέσουμε να άρουμε όλους αυτούς τους φραγμούς κατασκευαστικές βιομηχανίες, η, η, ο τομέας των ε, υπηρεσιών, οι δημιουργικοί τομείς υποφέρουν. Το ίδιο ισχύει και τους Ευρωπαίους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την πρόσβαση που θα ήθελαν σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο τέτοιων υπηρεσιών γιατί λιγότερο από το 10% του ευρωπαϊκού εμπορίου σήμερα ε, είναι διασυνοριακό ε, ακριβώ λόγω των συνδικών τη αγορά. Λιγότερο το 10% είναι διασυνοριακό από το ελληνικό εμπόριο. Επαναλαμβάνει ο μιλητή και ακόμα πιο ανησυχητική τάση σε σχέση με το τι γίνεται αλλού στον κόσμο είναι ότι δεν έχουμε διάβλους, δίκτυα διανομής. Ούτε πάροχους διαδικτύου που θα διένυμαν ψηφιακές υπηρεσίες. θα είμαστε εξαιρετημένοι από την ε, Αμερική. Αγοράζουν το βραγό περιεχόμενο οι Αμερικανοί και το διανέμουν πίσω στους Ευρωπαίους. Και επομένω, η υπεραξία, η αξία μάλλον μένει εκτός Ευρώπης. Και τους Ασιάτες το ίδιο ισχύει. Μιλάμε για εκατοντάδες δις ε, πελατών. Θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν ακριβώς το ίδιο δεν μπορείτε να βρείτε Ευρωπαίους παρόχους. Άρχιστε μια ματιά στις επικεφαλής του κλάδου. Από τα, από τα 50 πιο επισκέψιμα websites σε όλο τον κόσμο, στο διαδίκτυο, μόνο τέσσερα είναι ευρωπαϊκά. Επομένω, η Ευρώπη και στην κατάσταση κατά την οποία βαθμία ε, περιθωριοποιείται σε σχέση με τις ε, ε τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η ψηφιακή επανάσταση σε σχέση με την ε, βιομηχανία. Για δούμε τώρα ένα θέμα πιο συγκεκριμένο, το οποίο είναι από τα πιο επίμαχα, από τα πιο διφορούμενα και ε, έχει να κάνει με την, ε, με τη μη δημιουργία αγοράς. κανείς θα διαπιστώσει ότι τα δημιουργικά προϊόντα τα, τα αποτελέσματα των ε, δημιουργικών βιομηχανιών θα γίνουν ψηφιακά. Θα πρόκειται για την πρωτογενή διανομή του ψηφιοποιημένου περιεχομένου τα επόμενα χρόνια. Άρα σαν καταναλωτέ, όσο απολαμβάνουμε δηλαδή το αποτέλεσμα αυτών των δημιουργικών βιομηχανών, γίνεται μέσω του Ιντερνετ και μέσω αυτού του ψηφιοποιημένου περιεχομένου. Εάν δεν ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται σήμερα, στο διάστημα, να, να δούμε ας πούμε, τη, ε, μουσική βιομηχανία. Η, η ευρωπαϊκή ψηφιακή μουσική βιομηχανία είναι μόλις το τρίτον σε μέγεθος της αντίστοιχης αγοράς της Αμερικανικής. Πέρσι μεγάλωσε κατά 38% για ο αντίστοιχος τομέα στην Ευρώπη και στην Αμερική, ενώ λιγότερο από 10% ή στην, ε, Αμερική 38% και λιγότερο από 10% στην Ευρώπη. Επομένως, έχουμε αναλύσει εδώ και πολύ καιρό τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την μεταρρύθμιση στον ε, τομέα του copyright, ε, τους, οι αδειοδοτήσεις, ε, τα γεωγραφικά όρια, οι απαλλαγές και ο ρόλος των ενδιαμέσων. Επίσης, επανειλημμένα, έχουμε πει ότι χρειάζονται τρεις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη είναι τον έχουμε κάποιους καθιερωμένους μηχανισμούς για πιο αποτελεσματική, διαφανή ε, διαδικασία ε, αδειοδότησης για την διανομή του αυτού του ψηφιακού περιεχομένου. Αν δούμε ακριβώς τα, τη διαχείριση, ώστε να μπορούν οι εμπλεκόμενοι με τρόπο εύκολο αλλά και διάφανο να, να δουλέψουν, τόσο ώστε να έχουμε μια καλύτερη ε, διανομή στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ε, δασμούς όσον αφορά ε, το copyright και αυτό είναι ένα πρόβλημα και επίσης υπάρχει κατάτμιση στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν ανταποκρίνονται αυτές τις ανάγκες της ε, ψυχικής εποχής. Private copy. Τι είναι αυτό. Θα πρέπει κάπου αυτό το ιδιωτικό αντίγραφο να οριστεί. τι θα πει εύλογη και δίκαιη αποζημίωση. Προβλέπεται αυτό στο δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για το τι είναι τέτοια δίκαιη αποζημίωση παρά το ότι στο δίκαιο προβλέπεται ότι η αποζημίωση εξαρτάται από την πραγματική ζημία που υπέστη ο δημιουργός. Εάν λοιπόν αυτό το δίκαιο της πραγματικής διοκτησίας ε, μεταρρυθμιστεί, αυτό θα βοηθήσει και τη βιομηχανία γενικότερα. Κατά τρίτο λόγο επίσης χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση όσον αφορά την διακυβέρνηση σε σχέση με τους ενδιάμεσους. Αυτές οι εισπρακτικές εταιρείε του ΣΥΠΗΝ δεν υπάρχει εκεί πέρα διαφάνεια, δεν υπάρχει λογοδοσία με τον συμβατικό τρόπο όπως ακριβώς γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τις εταιρείες σε σχέση με τη χρήση των χρημάτων. Γιατί υπάρχουν κάποια είδους ε, παραδείγματα όπου είναι δυνατόν αφού εισπραχθεί το εισόδημα να πληρωθεί ο καλλιτέχνης πέντε χρόνια αργότερα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, που πάρα πολλοί θα δικαιούνται το σχετικό εισόδημα και δεν παίρνουν ποτέ τα λεφτά που πρέπει. Και υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων Οπότε οι καλλιτέχνε δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην αγορά γιατί δεν θέλουν αξιόπιστοι παίκτε από αυτού του ενδιαμέσου. Επομένω, έχουμε αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Είναι τα θεμέλια τα που χρειάζονται για να φτιάξουμε αυτήν την ενιαία αγορά. Άρα θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Βλέπουμε τη σημερινή τάση που οδηγεί στην περιθωριοποίηση τη Ευρώπη Χάνονται οι ευκαιρίε που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση. Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτοί που πάνε σε Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβούν στι αναγκαίε μεταρρυθμίσει, ώστε να έχουμε οικονομική ευημερία και, και κοινωνική ευημερία για όλου του Ευρωπαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Όρμαλα. Μας τρόμαξαν αυτά που είπατε, τουλάχιστον εμένα. Ε, ελπίζω να έχουμε καλή σύντηση που θα ακολουθήσει. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πουαρό, ιδρυτή του European Cinemas. Ευχαριστώ. Θα ήθελα στην αρχή, από την αρχή να πω κάτι για τις πρώτες δημοσιεύσεις του κυρίου Πιότρ Μπορίση για, το, για τα ψηφιακά. Τα εκτιμήσαμε ιδιαιτέρως. Εγώ θα πω μερικά πράγματα πιο περιορισμένου εύρους. Τέσσερα κύρια σχόλια έχω να κάνω. Το ενδιαφέρον και η αναγκαιότητα να εξοπλιστούμε ψηφιακά ο κατεπήγον χαρακτήρας του εξοπλισμού αυτού, οι ανισότητες μεταξύ των αιθουσών ως προς τα ψηφιακά και οι προοπτικές του ψηφιακού για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Πρώτον, το ενδιαφέρον και η αναγκαιότητα να εξοπλιστούμε. Μετά τον ήχο, τα ειδικά εφέ, το ίδιο το γύρισμα, η προβολή η ίδια γίνεται ψηφιακά και σιγά σιγά αντικαθίστανται οι μηχανές των 35 mm που επί έναν αιώνα ήταν εκείνες που κυριαρχούσαν για την προβολή των έργων παγκοσμίω. Εξού η αναγκαιότητα σήμερα να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο ασφαλές σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα που να το εγκρίνουν και να το δεχτούν όλοι οι εκπρόσωποι του τομέα, οι επαγγελματίες. Τώρα για τον θεατή. Ο θεατής είναι όλο και πιο απαιτητικό γιατί ήδη και στο σπίτι του χρησιμοποιεί πολύπλοκες μηχανές. Η ψηφιακή προβολή στην αίθουσα του δίνει την ασφάλεια να δει σε μεγάλες οθόνες μια εξαιρετική εικόνα η οποία δεν χαλάει καθ' τη διάρκεια ζωής του έργου και του δίνει πρόσβαση και στις τρεις διαστάσεις που δίνουν μία νέα προοπτική. Μετά από τον James Cameron και τον Wim Wenders και άλλοι Ευρωπαίοι κινηματογραφιστέ ενδιαφέρονται στη στερεοσκοπία. Τέλος για τον ε, ιδιοκτήτη της αιθούσης. Μπορεί να λαμβάνει τα έργα σε πιο ελαφριά μορφή, να μην χρειάζεται τεράστια αποθήκευση, μεταφορά, καταστροφή το, της κόπιας κλπ. Και μπορεί επίσης να διαφοροποιήσει την προσφορά του και σε άλλου είδους περιεχόμενα να προβάλλει κατευθείαν ανεμεταδόσεις όπερας ή άλλα. Και επίσης θα μπορεί να διατηρεί στη βιβλιοθήκη του τους τίτλους και να τα ξαναπέζει όποτε θέλει εκείνος ή το κοινό ή για ειδικέ περιστάσεις όπως για σχολικές προβολές. Δεύτερον, ότι είναι επίγον να εξοπλιστούμε. Σε πολύ λίγα χρόνια ο ολόκληρος ο τομέας του σινεμά εξοπλίστηκε ψηφιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Κίνα. Οι υπάρχουσες αίθουσες παράτησαν πια τις μηχανές των 35 χιλιοστών και δέχτηκαν αυτή τη νέα τεχνολογία. Οι δε καινούργιε αίθουσε κατευθείαν είναι εξοπλισμένε για το ψηφιακό χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου τα 35 χιλιοστά. Είναι σχεδόν ε, παγκόσμιο το πρότυπο αυτό πια. Η Ευρώπη στο σύνολο των κινηματογράφων της έχει ψηφιακές οθόνες για την προβολή έργων τρισδιάστατων και οι ιδιοκτήτες ζητούν ε, ψηφιακές κόπιες. Για να μην υπλασιάσουν τα έξοδά τους, οι διανομής είναι πρόθυμοι να διαθέσουν κατευθείαν ψηφιακές κόπιες που είναι 5 με 10 φορές λιγότερο ακριβές. Μια αίθουσα που σήμερα θα περιοριζόταν στις μηχανές 35 χιλιοστών αναλαμβάνει τον κίνδυνο να κλείσει μέσα στους επόμενους μήνες γιατί δεν θα τροφοδοτείτε πια από τους διανομής που δεν διανέμουν παραδοσιακά φιλμ. Για αυτούς τους τεχνικούς και οικονομικούς λόγους το σύνολο του τομέα θα ήθελε να επιταχύνει αυτήν την ε, αλλαγή. Όσοι αργήσουν θα ζημιωθούν βαριά. Τρίτο θέμα, οι διαφορές των αιθουσών. Στην Ευρώπη 1.130 αίθουσες αντιπροσωπεύουν 35% των οθονών με πολύ προωθημένη ψηφιακή εγκατάσταση. Οι άλλες, οι άλλες έχουν διαφορετικά για τις άλλες ισχύουν διαφορετικά στοιχεία. Για την πρώτη προβολή, συχνά πολυέθουσε με γιγαντοοθόνες, υπάρχουν σε καμιά δεκαριά μεγάλες χώρες, και μπορούν εκεί οι ιδιοκτήτες άμεσα ή έμεσα χάρη σε τρίτους να πάρουν από τους διανομής ε, ορισμένα χρήματα γιατί εξοικονομούν με σύγκριση, σε σύγκριση με την παραδοσιακή κόπια. Αυτό το σύστημα που λέγεται VPF είναι μια λύση για την αυτοχρηματοδότηση των αιθουσών Σχεδόν οι μισές από τις 815 αίθουσες του δικτύου Europa Cinema ε, είναι αυτού του τύπου. Δυστυχώς στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές μικρές αγορές όπου ο αριθμός που κυκλοφορεί των κοπιών είναι πολύ ανεπαρκής για να χρηματοδοτήσει τις νέες εγκαταστάσεις. Γιατί σας υπενθυμίζω 80.000 ευρώ χρειάζονται ένα αίθουσα. Υπάρχουν και πολλές μικρές αίθουσες με μία ή δύο οθόνες που είναι πάρα πολλές στις μικρές και μεσαίες πόλεις της Ευρώπης αλλά που δεν έχουν τα μέσα να εγκαταστήσουν τα νέα μηχανήματα. Ο κίνδυνος είναι αυτές να χρειαστεί να κλείσουν ενώ έχουν λόγο ύπαρξη στην αγορά και κοινωνική ζωή στην οποία συνεισφέρουν. Εκτός αν δημόσια μέσα και πόροι, ευρωπαϊκά, εθνικά ή περιφερειακά, συμπληρώσουν τους πόρους της αγοράς. Στο δίκτυο Europa Cinemas που έχει 2.000 ε, οθόνες ευρωπαϊκού κυρίως προγραμματισμού υπάρχει ο κίνδυνος να εξαφανιστούν μερικές εκατοντάδες αίθουσες που σήμερα αποτελούν τον πλούτο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι επίγον και απαραίτητο να βοηθήσουμε τις αίθουσες αυτές να εξοπλιστούν και να συνεχίσουν την πολιτιστική και κοινωνική αποστολή τους. Σε μερικές χώρες όπως τη Γαλλία, την Ορβηγία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα. Άλλα, άλλες χορηγούν βοήθειες σε ορισμένα είδη αιθουσών. Αυτές οι πρωτοβουλίες δυστυχώς δεν αρκούν και αφήνουν ε, και είναι και άνηση η διανομή του στην Ευρώπη. Αφήνει πολλές αίθουσε χωρίς πόρους, ενώ είναι θεμητή η ύπαρξή τους. Το πρόγραμμα Μίδια και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ήδη σε θέση να βοηθήσουν. Αλλά τονίζω ότι πρέπει να προσέξουμε τι, το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει κάτι επίγον εδώ. Τέλος, η προοπτική του ψηφιακού για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Η ψηφιακή προβολή δίνει στις αίθουσες τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν την προσφορά τους. Το λιγότερο κόστος εξόδου ενός έργου, οι πολλές, πολλαπλές δυνατότητες υποτίτλων και ντουμπλάζ δίνουν σε όλους δυνατότητες που δεν είχαν προηγουμένως ιδιαίτερα στις μικρότερες αγορές. Αν παράγονται, θα μπορούν έτσι να παράγονται περισσότερα έργα στην Ευρώπη και να κυκλοφορούν με καλύτερες συνθήκες οι ευρωπαϊκές αίθουσες. Αυτό είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους οι αίθουσες και για να φτάσουν πιο κοντά στο κοινό τους τα ευρωπαϊκά έργα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποικιλομορφία είναι βασικό στοιχείο των ανεξαρτήτων αιθουσών. Εξάλλου αυτή η ιστορική μεταβολή στις αίθουσε θα συνδυαστεί με την εξέλιξη των μέσων προώθησης, δηλαδή οι αίθουσε στο δίκτυό μας τουλάχιστον ήδη το έχουν κάνει αυτό χρησιμοποιώντας ό,τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν από αυτήν την ε, ψηφιακή επανάσταση, δηλαδή την ανακοινώσει με ίντερνετ, τα blog και τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η τεχνολογική πολιτική περιπέτεια είναι διαδραστική και δίνει μεγάλες ευκαιρίες στις αίθουσές μας να παίξουν ένα ρόλο επιμορφωτικό για τους νέους ιδιαίτερα. Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι στη γλώσσα των εικόνων σημαίνει να του συνηθίσουμε να προτιμούν τα ευρωπαϊκά έργα, αυτά που βλέπουμε στα φεστιβάλ. Στην Ευρώπη έχουμε σκηνοθέτες τεράστιου ταλέντου και μεγάλης φήμης και επίσης έναν αριθμό αιθουσών εξαιρετικό. Το ψηφιακό λοιπόν πρέπει να τους βοηθήσει και τους μεν και τους δε έτσι ώστε η κινηματογραφική αίθουσα να παραμείνει αυτή που πάντα ήταν δηλαδή ένας μοναδικός τόπος συνάντησης και πολιτισμού προσβάσιμος σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Äh, και τώρα έχουμε τον ε, Γενικό Γραμματέα της ΕΓΕΝΤΑ, ο κύριος Σουάρες Λουτσάνο, ο οποίος καταρχήν μπορεί να μας πει τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΓΕΝΤΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε την οργάνωση που εκπροσωπώ και ακολουθώντας ε, το παράδειγμα του Ιταλού ε, συναντέλφου θα μιλήσω και εγώ ισπανικά. Η Έγκεντα είναι μια εταιρεία η οποία εκπροσωπεί τους ε, παραγωγούς ε, οπτικοακουστικών παραγωγών στη Γαλλία. Δηλαδή εκπροσωπούμε πάνω από 1.400 παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και λατινοαμερικανοί καλλιτέχνες, οι οποίοι βέβαια για πάρα πολλούς λόγους είναι στενά συνδεδεμένοι με την Ισπανία. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχει ε, σαφής ε, διαχωρισμός, διότι στον οπτικοακουστικό τομέα το οικονομικό μοντέλο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στον τομέα της ε, μουσικής και τα νομοθετικά εργαλεία δεν μπορούν να είναι ίδια. Το σύστημα η ύπαρξη ενός συστήματος ε, εκμετάλλευσης της μουσικής είναι ένα παράδειγμα. Και ε, όταν ε, δραστηριοποιούμε τα νομοθετικά, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα, οι νόμοι είναι εκείνοι που καθορίζουν το οικονομικό μοντέλο και το οπτικό-ακουστικό μοντέλο. Είναι λοιπόν σαφές ότι αν αλλάξουμε το μοντέλο, τότε αυτό θα είναι ένα άλμα στο κενό. Ε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ε, μπορεί να προκύψει. Όσον αφορά τώρα στον οπτικοακουστικό τομέα, όπως σας είπα, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε το ρόλο των εταιριών παραγωγής στον οπτικοακουστικό τομέα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Ε, αυτή τη στιγμή ε, είμαστε περιοριζόμεθα στα ιδιωτικά αντίγραφα όπου υπάρχουν αυτά ε, και στην μετάδοση, την καλωδιακή. Οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης δεν είναι αποδεκτή. Ας δούμε τώρα οι εταιρείε διανομής τι ρόλο η εκμετάλλευση, τι ρόλο μπορούν να παίξουν. Πρώτον, πρέπει να δούμε τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά να τα εξετάσουμε κάτω από το πρίσμα του παραγωγού. Οι μηχανισμοί της αγοράς δεν αρκούν ε, για να διασφαλίσουμε ε, την πρόσβαση των πολιτών σε ένα μεγάλο κομμάτι των οπτικοακουστικών έργων. Είναι λοιπόν απαραίτητο η εσωτερική αγορά να ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης. Ε, εδώ μιλάμε για μεγάλους ε, καταλόγους και μιλάμε κυρίως για τους Αμερικανούς οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλη ζήτηση. Έχουμε και τα επίκαιρα έργα στην Ευρώπη, ε, τα οποία ε, σημείωσαν επιτυχία και κατά το παρελθόν. Μια άλλη πραγματικότητα που καλούμετα να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη κοινή γλώσσας. Και αυτό σημαίνει ότι προκύπτει επιπρόσθετο κόστος. Βεβαίως αυτό έχει επιπτώσεις ε, στη ζήτηση και επιπλέον κάτι τέτοιο περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά, κυρίως όταν πρόκειται για ανεξάρτητους παραγωγούς. Ας δούμε τώρα ποια είναι η εναλλεκτική λύση για εκείνους που αποκλείονται. Η ατομική ή ομαδική πρόσβαση στην αγορά ή σε μικρές αγορές εξειδικευμένες που υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη. Αυτό όμως σημαίνει ιδιαίτερα υψηλό κόστος για ανεξάρτητους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών. Κόστος υποδομής, η απαραίτητη ευρυζωνικότητα για να είναι κανείς ανταγωνιστός και το κόστος συναλλαγής στις πληρωμές. Αυτό το κόστος μερικές φορές είναι και μέχρι το 50% ανάλογα με το ποιο μέσο πληρωμής χρησιμοποιούμε. Ανάλογα με το τι κεκτημένο υπάρχει επομένω στην Ευρώπη για τα οπτικοακουστικά, επομένω η συνέπεια είναι ότι εκείνε παραγωγέ που δεν φτάνουν στην αγορά ε, ό, όταν ε, αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν υπάρχει ζήτηση και τελικά δεν υπάρχει ούτε προσφορά, λιγότερη προσφορά ευρωπαϊκή και συγκεκριμένα υπάρχει μια διαφορετική, διαφοροποιημένη προσφορά. Οπότε, με δεδομένη αυτή την κατάσταση που έτσι πάει να γίνει, τότε ε, μετακυλείται το θέμα στον ε, δημόσιο τομέα και έτσι βλέπουμε τι είδους μηχανισμοί υπάρχουν για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην, στην αγορά. Και αυτό πώς γίνεται μόνο με την επιδότηση, με τη στήριξη από το δημόσιο. Επίσης, ε, ε, αυτές οι εταιρείες της διαχείρισης τελικά είναι ο καταλήτης. Και αυτό γιατί, γιατί έχουν ε, άμεση επαφή, έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, πρόσβαση στην πραγματικότητα στην Ισπανία. Έχουμε μία πύλη με παραγωγούς Ισπανίων από, από το 2006, από το Μάη του 2006. Αυτό άνοιξε προς όλη την Ευρώπη και είναι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να εισφέρουμε ως δική μας ε, και χτυμένη εμπειρία. Έχουμε περίπου 900 ε, τίτλους που έχουν ανέβει στο ίντερνετ και αλλιώς χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε κανεί να έχει πρόσβαση να, τις, να δει αυτέ τι ταινίε. Οπότε για να υπάρχει τελικά μια ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά η οποία να είναι ισχυρή εύρωστη θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιβάλλον νομοθετικό κατάλληλο, πρόσφορο. Και επομένω ένα από τα πρώτα βήματα είναι το να ενημερώσουμε την οδηγία 48 του 2004. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να γυρίζουμε την πλάτη στη πραγματικότητα που για πολλές χώρες ε, οδήγησαν σε καταδίκες από το, από, από δικαστικές όπως αυτό προήλθε από σύγκρουση με τις εταιρείε διαχείρισης ιδιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και οπότε αυτοί οι οποίοι είχαν ε, παραβεί το δίκαιο ε, υπέστησαν τις κυρώσεις. Ε, επομένως, χρειάζεται να υπάρχει και το κατάλληλο πλαίσιο και επίσης για μας, για τη διαχείριση, θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των ορφανών δημιουργημάτων, έργων. Κατά τη γνώμη μας, το σχέδιο της οδηγίας, το οποίο τώρα επεξεργάζεται η Ένωση, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά ε, οπωσδήποτε επιδέχεται βελτίωση αυτή η κατάσταση πρώτα-πρώτα γιατί δεν υπάρχει αρκετή μελέτη του προβλήματος γιατί ε, δεν ξέρουμε καν πώς είναι τα ορφανά έργα στην Ευρώπη. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση ε, στις Mediatek, στις φιλμοθήκες ε, ε, όπου δεν κατατίθενται τα έργα. Εκεί κατατίθενται αντίγραφα των έργων που είναι κινητά πράγματα και επομένως γίνονται αντικείμενα σύμβαση παρακαταθήκη σύμφωνα με τον αστικό κώδικα και οπότε μετά υπάρχουν προβλήματα για να, να επισημανθεί, να βεβαιωθεί, να σιγουρευτεί η κυριότητα αυτών των κινητών ε, αγαθών. Και επίσης ε, υπάρχει πρόβλημα και με τους καταναλωτές για αυτά τα έργα και το σχέδιο της οδηγίας έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης αυτών και ήδη αυτά έχουν ανατεθεί ε, σε κάποιες εταιρείες διαχείρισης που όμως κάποιες έχουν, έχουν εξαφανιστεί και επομένως το, τα, τα προγνωστικά για την ε, για το διαχείριση είναι 27 διαφορετικές λύσεις που θα υπάρχουν στα επόμενα 2-3 χρόνια εάν δεν ε, βιαστούμε την οδηγία αυτή να την μεταφέρουμε στο εσωτερικό δίκαιο και δεν έχουμε δηλαδή αντιδράσει με την ταχύτητα που απαιτείται από πλευράς του κοινού. Ε, γιατί υπάρχει όντω τέτοια απέτηση, τέτοια ζήτηση από πλευρά του κοινού. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις εταιρείε διαχείριση. Φυσικά και μπορούν αυτές κάτι να κάνουν για τα ορφανά έργα. Ε, έχουν τι πληροφορίε όσον αφορά τους δικαιούχου και επομένως μπορεί να γίνει μια ευφυή αναζήτηση, έχουν την ε, εμπειρία, μεγάλους καταλόγους να τους ε, διαχειρίζονται και επίσης ε, ξέρουν να κινούνται για τις κατάλληλες, ε, τιμέ τιμές για τις συναλλαγές και αλλιώς κινδυνεύει κανείς να καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια όπως ήδη έχει γίνει και κατά αυτόν τον τρόπο θα, υπάρχει και δημόσιος έλεγχος και διαφάνεια. Αυτές οι εταιρείε επίσης έχουν κάποια σταθερότητα στην πορεία τους μέσα στον χρόνο και επίσης ε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά με λιγότερα έξοδα από όσο το δημόσιο. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτές οι εταιρείε είναι η απάντηση στο πρόβλημά μας, το κατάλληλο εργαλείο για να λύσουν το πρόβλημα. Επίσης, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κάποια στιγμή να δούμε πώς θα ρυθμιστεί η πνευματική ιδιοκτησία σε μία ενιαία αγορά. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία αγορά με 27 διαφορετικές νομοθεσίες. Χρειάζεται κάτι το οποίο προοδευτικά μας εμποδίζει περισσότερο, λένε, και περισσότερο, δεν ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Οπότε, από πλευρά Ισπανών παραγωγών θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Ε, οι οδηγίες μέχρι τώρα έχουν βοηθήσει. Ήταν μια χαρά νομοθετήματα. Όμως, τη σήμερα ημέρα έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο η οδηγία, η ερμηνεία, συγγνώμη, θα πρέπει να γίνεται από το δικαστήριο ή τα δικαστήρια. γιατί εκτός από τις ε, αποφάσεις των σημάτων δεν περνάει τρίμηνο χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους ε, αποφάσεις. Άρα χρειάζεται κάποιο είδους νομοθεσία, κάποιο είδους ρύθμιση που να μας δώσει την απαραίτητη ανταγωνιστικότητα. Με του ανταγωνιστέ μα δεν θα πρέπει να αναμετρηθούμε γιατί αυτοί έχουν αυτά τα μέσα που σα είπα στη διάθεσή του. Και ενώ η αγορά του είναι όπω η δική μα. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Όλα αυτά που ακούσαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, έδωσαν τροφή στη δουλειά μας, τη δουλειά που θα έχουμε κατά τους επόμενους μήνες. Ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, την κυρία Τρούιπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντόρις. Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω αυτές τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που ακούστηκαν και να υποβάλω τις ερωτήσεις μου. Γιατί προέβαλαν ε, διαφορετική διάσταση των πραγμάτων με διαφορετικό υπόβαθρο. Ε, εκείνο που κατανοώ πολύ καλά είναι ότι επιθυμούμε να υπάρξει ψηφιακή κοινή αγορά. Όμως το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και με ποιους κανονισμούς διότι προφανώς, ε, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, αν δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχει και μεγάλος ε, κίνδυνος. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε ψηφιακή κοινή αγορά, γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να καταλήξω τώρα σε κάποιες ε, έντονες ε, αντιφάσεις που υπάρχουν εδώ και τρία χρόνια. Στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο άρθρο 27, γίνεται λόγος για την ελεύθερη πρόσβαση στην ε, πολιτιστική κληρονομιά και στο ίδιο άρθρο έχουμε και την προστασία του copyright. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι πρέπει να καλύψουμε και τους δύο στόχους και τώρα φτάνω στις ε, ερωτήσεις μου, γιατί ελπίζω να μπορείτε να μου δώσετε κάποιες ε, απαντήσεις. Ε, Ξεκινώ με τον πρώτο μιλητή που είπε ότι, είμαστε ναι, που είπε ότι ναι, είμαστε υπέρ της ουδετερότητας, αλλά επιθυμούμε τη διαφάνεια των όσων συμμετέχουν στο διαδίκτυο ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα είδους ε, ευθύνης ε, που αναλαμβάνουν οι χορηγεί στο, οι φορείς που παρεμβαίνουν στο διαδίκτυο ευθύνη ως προς το τι κάνουν με τα δεδομένα, τι γίνεται με τον ορισμό του εμπορικού και του μη εμπορικού. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναφερθήκατε σε ε, διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας ε, για όλους. Αλλά ποιος θα το πληρώσει αυτό, το κράτος. Οι άνθρωποι ε, αν δεν έχουν τα χρήματα για διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας τότε ποιος θα πληρώσει αυτή την ταχεία πρόσβαση. Κατόπιν μιλάτε για ευρωπαϊκό ψηφιακό διαβατήριο. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό. Και πάω τώρα στον ε, εκπρόσωπο ε, της Nokia. Εσείς ως εταιρεία Nokia είναι σαφές το ότι επιθυμείτε ε, να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο, όσο δυνατόν περισσότερο την ψηφιακή αγορά της Ευρώπης. Και μιλάτε για μεταρρύθμιση και θα ήθελα ε, να ενημερωθώ λιγάκι για τους ε, ορισμούς σας. Λέτε πρέπει να ορίσουμε τι είναι το ιδιωτικό αντίγραφο. Ε, παλαιότερα οι φίλοι σας να, μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιωτικά αντίγραφα. Τώρα όμως πλέον τίποτα δεν είναι ιδιωτικό και μπορεί κανείς να μοιραστεί το ίδιο αντίγραφο με εκατομμύρια ανθρώπων. Τι ακριβώς σημαίνει ιδιωτικό αντίγραφο σε ψηφιακό περιβάλλον. Τι ορισμό δίνεται. Δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε για συλλογική αδειοδότηση, ε, κανένα πρόβλημα και κατόπιν μιλάτε για δίκαιη αποζημίωση. Τι είναι ακριβώς αυτή η δίκαιη αποζημίωση. Είναι ένα καταποκοπή ποσό, είναι ένα ποσό ε, που αφορά τις εισφορές επιβάλλεται νομικά υπάρχει δυνατότητα του opting out υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα σχετικά με τη δίκαιη αποζημίωση και τι ακριβώς γίνεται τελικά είναι η λύση της αγοράς, είναι η λύση του κράτους αυτά δεν μου είναι απόλυτα σαφή Κατόπιν μιλάτε για τις ε, μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ όπως είναι η Google που ε, εκμεταλλεύονται και κερδίζουν από το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ε, και τι γίνεται όμως με τους καλλιτέχνες αμείβονται σωστά. Εγώ δεν είμαι κατά νέων επιχειρησιακών μοντέλων αλλά τι ακριβώς ε, συνεπάγονται αυτά ε, για τους ε, καλλιτέχνες. Μπορούν να ζήσουν από τα χρήματα αυτά. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για το ψηφιακό περιβάλλον. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του copyright, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε και οι καλλιτέχνες να βρίσκονται σε καλύτερη θέση όσον αφορά τους νέους φορείς που συμμετέχουν στο διαδίκτυο. Ελπίζω να τα θυμάστε όλα αυτά, όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω πόσο ενδιαφέρον είναι εμείς οι Ευρωπαίοι ε, με τη βοήθεια των ε, εμπλεκομένων στον κλάδο ε, των δημιουργών να, να, να, να ενημερωνόμαστε γιατί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό ε, πρόκειται για ένα τομέα όπου έχουμε δυνατότητες, έχουμε αδυναμίες και δεν είμαστε τόσο καλά οργανωμένοι και το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει περιορισμός της υποδομής, της βιομηχανίας, της πολιτιστικής, ε, της σύλληψης των δυνατήτων μας και επίσης θα ήθελα να σας πω το, το, εξής και, και συγγνώμη πρέπει να φύγω ότι έχουμε στην Επιτροπή μας να ζητησουμε έναν Επίτροπο πρώτα πρώτα όσον αφορά το, το, το, το, το ψηφιακό σύμπαν νομίζω ότι ε, θα πρέπει, ε, ξέρουμε τώρα οι πιο βασικοί παράγοντες ε, συμφωνούν ότι τώρα έχουμε την τρίτη επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είχαμε πρώτα-πρώτα την επανάσταση στη Γεωργία και όταν βρέθηκαν τα δικά εργαλεία, μετά τη βιομηχανική και τώρα έχουμε αυτό το, το, το σήμα και είναι μια τρίτη επανάσταση. Περί πρόκειται, είναι μια επανάσταση η οποία ε, για άλλη μια φορά όπως οι άλλες δύο επαναστάσεις έρχονται μέσω του εργαλείου και το εργαλείο βέβαια είναι το ψηφιακό εργαλείο ε, και υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα τα οποία έθιξαν οι προσκεκλημένοι μας και εγώ θέλω να σταθώ σε ένα ότι έχει μεγάλη δυσκολία η Ευρώπη δεν μπόρεσε παρά τα χρήματα που υπάρχουν δεν μπόρεσε να φτάσει ε, σε, σε μια διείσδυση της ψυχικής τεχνολογίας παντού και στην, και στην Ήπεθρο ακόμα. Και θα πρέπει να υπάρχει πολιτισμός, να υπάρχει αποζημίωση, αμοιβή, ικανή, ικανοποιητική σε αυτούς που δημιουργούν και σε αυτούς που διανέμουν. Επίσης κάτι άλλο για την τηλεόραση. Ε, θα ήθελα να μου πούνε εδώ ήρθε και ο συνάδελφος και φίλος Ιγνάση Γκορντάνς ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί αυτό το οποίο τώρα με εντυπωσιάζει είναι ότι σιγά σιγά η Ευρώπη στο όνομα ε, αυτού του ε, ιερού και όσου του, του ανταγωνισμού του 1980 ε, χάθηκε ε, αυτό το, το ισορροπημένο το οποίο που υπήρχε ε, και υπήρχε ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημοσίων και ο καθένας παρήχε στον τομέα του διαφορετικά πράγματα και μετά ε, η στον τηλεθεατή ανάλογα με το τι προτιμάει. Επίσης θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον εκπρόσωπο ε, της ε, ΙΕΡ και ε, όσον αφορά την παραγωγή κάποιων έργων που είναι κάτι παραπάνω, κάτι παραπέρα από τα τηλεπαιχνίδια και επίσης νομίζω ότι η υπηρεσία πληροφόρησης είναι πάρα πολύ βασική είναι κάτι στο, το οποίο έχει να κάνει και με τι, κάτι, κάτι το οποίο λείπει σε πολλές χώρες. Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Οπότε, έτσι νομίζω ότι θα, θα, ε, θα ο κόσμος, θα ελκυστεί να τα ακούει και επίσης κάτι άλλο, η χρήση της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου με οποιαδήποτε τεχνολογία. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει ανεξαρτησία και σταθερότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση εξαρτησία σε σχέση με την πολιτική εξουσία. Δεν θα σας πω σε ποιες χώρες για να μην ε, στεναχωρηθεί κανένας, αλλά ε, δεν, σε χώρες κεντρικής Ευρώπης δεν συμβαίνει αυτό. Στις δημόσιες επιχειρήσεις και θα πρέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να το προσέξει. Έχουμε κάποια προγράμματα διασκέδαση, προγράμματα, προγράμματα εκπομπέ γνώση, ε, ιστορικέ εκπομπέ, γενικής ενημέρωσης που θα πρέπει να μπορεί κανείς να τα δει, να τα ακούσει ε, με διαφορετικές τεχνολογίες. Και αυτό γιατί οι νέες γενιές φεύγουν από την Ατζιανή, τηλεόραση Ατζιανή μετάδοση και ε, αυτή ακριβώς είναι εκείνη που τους λείπει αυτή η ενημέρωση. Εκεί, αυτή, ε, εκεί χρειάζεται η δημοκρατική ενημέρωση. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη, περισσότερο από ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Καβδά και τώρα... Ρόχιο Μπόρις ο συγκεκριτής. Ε, ευχαριστούμε για θα ήθελα όμως να θέσω και ένα ερώτημα στους εμπειρογνώμονες. Από τη μία, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η προσφορά, η πολιτιστική προσφορά να επεκταθεί η οπτικοακουστική προσφορά στους Ευρωπαίους καταναλωτές και καταναλώτριες. Να εφαρμοστεί η σύμβαση που ανέφερε η κυρία Τρούπελ. Απ' την άλλη Ξέρουμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν μεγαλύτερες δυνατότητες για τη βιομηχανία. Θα υπάρχει καλύτερη πρόσβαση δηλαδή. Και αυτό φαίνεται ήδη από την Αμερικανική αγαρά. έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών εμείς στην Ευρώπη και αυτό θα αυξήσει και τα εισοδήματα. Έχω όμως το ερώτημα πώς μπορούμε χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και οι καινούργιες γενιές που ήδη χρησιμοποιούν ε, μη γραμμικές υπηρεσίες και άρα θα αυξηθεί η ζήτησή τους. Πώς από τη μία λοιπόν διασφαλίζουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την δίκαια αποζημίωση των δημιουργών και από την και απ' την άλλη πώς θα διασφαλίσουμε ταυτόχρονα οι καταναλωτές και καταναλώτριες να αποφεύγουν την παράνομη χρήση. Γιατί ξέρουμε ότι είναι τεράστια η παράνομη αγορά στην Ευρώπη. Νομίζετε, θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και η καταναλώτρια σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποτελεσματικά αλλά χωρίς παρανομία. Χωρίς παρανομία. Ευχαριστούμε κύριε Καμέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τους τέσσερις ομιλητές. Ο κύριος Ματσόνε μας αποσαφήνισε ακόμη μια φορά ότι η καλύτερη τεχνολογία αν δεν έχει κάποιο περιεχόμενο να προσφέρει είναι τελείως άχρηστη. Μιλάμε για ψηφιοποίηση και τεχνολογία αλλά ξεχνάμε ότι χρειάζεται και περιεχόμενο για όλα αυτά. Αυτό είναι ουσιώδες. Και είναι κάτι που πρέπει να το λέμε συνεχώς. Μιλήσαμε για ουδετερότητα του δικτύου, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Κομισιόν καθυστερεί, διστάζει να νομοθετήσει για την εγγύηση των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, αλλά εσείς τι φρονείτε, χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη ώστε να μην υπάρχει άνηση μεταχείριση για το περιεχόμενο διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το κλασικό περιεχόμενο αλλά υπάρχουν και τα δίκτυα που προσφέρουν παράνομα ή δωρεάν ανάλογο περιεχόμενο πρέπει να επιλέξουμε ορισμένα είδη περιεχομένου με δικαιώματα και άλλο είδος χωρίς δικαιώματα. Επίσης πρόσφατα είδαμε, ανακάλυψα ότι υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες υβριδικές τηλεοράσεις. Οι Ιταλοί επέλεξαν ένα σύστημα που λειτουργούν με διάφορα συστήματα δηλαδή, γιατί άλλο είναι το Ιταλικό, άλλο το Γερμανικό μήπως χρειάζεται κάποιο είδος ευρωπαϊκής τυποποίησης γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού αν οι κατασκευαστές δηλαδή αντιμετωπίσουν δυσκολίες γιατί είναι μικρή η παραγωγή τους λόγω του συστήματος που χρησιμοποιούν σε σύγκριση με άλλους κλπ. Ίσως λοιπόν εδώ η ευρωπαϊκή τυποποίηση να ήταν κάτι το θετικό τέταρτον για τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright δηλαδή. Μου αρέσει η ιδέα αυτού του ιδιωτικού αντιτύπου. Αλλά αναρωτιέμαι αν έχετε και εσείς καμία ιδέα ως προς το πώς θα μπορούσε αυτή η ιδέα να μεταφερθεί στον ψηφιακό κόσμο ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ των δικαιωμάτων των δημιουργών από τη μία και της δυνατότητας του κόσμου να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο από την άλλη. Να μας πείτε μερικά λογάκια. Αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου κύριο μου, η κυρία Κώστα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για την απόφαση που έλαβε να προχωρήσουμε σε αυτή την ακρόαση που είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Κυρίως γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση ιδιαίτερα περίπλοκη και υπάρχουν θέματα εδώ που δεν αφορούν μόνο από την Επιτροπή αλλά και άλλες επιτροπές. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι το θέμα της ψηφιοποίησης, ε, της παραγωγής, ε, της ε, Βιομηχανική οικονομίας και του πολιτισμού. Ε, όλα αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερης ε, σημασίας ε, και το είπα νομίζω αυτό και προηγουμένως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν το λόγο για την σαφήνεια με την οποία μίλησαν και για τις προτάσεις που έκαναν. Και όσον αφορά την παρέμβαση του κυρίου Ματσόνε, νομίζω είναι σαφές και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ε, ότι υπάρχει στην Ευρώπη ένα διτό σύστημα, αλλά το πρόβλημα κατά κύριο λόγο είναι το εξής. Και το λέω μία και μόνο πρόταση. Οι πόροι που αφορούν την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη μεταφέρονται από τα οπτικοακουστικά, από όριμες ε, βιομηχανίες αν θέλετε, μεταφέρονται ε, στα δίκτυα, στα ψηφιακά προϊόντα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε όλη αυτή την αλυσίδα αξιών. Και αυτό θέτει ένα μεγάλο ερώτημα. Με ποιους κανόνες θα γίνουν όλα αυτά και προς ποια κατεύθυνση. Η Ευρώπη θέλει να προτείνει με τις επόμενες οδηγίες ότι δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας κάτι το σημαντικό. Ότι οι επενδύσεις σε ποιοτικέ παραγωγές, ε, ε, οι εγγυήσεις που προσφέρονται στους πολίτες, όλα αυτά ε, προέρχονται από κρατικά κανάλια και υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τα κρατικά κανάλια. Αυτά δεν είναι παρόντα μόνο στην ψηφιακή παραγωγή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ο, η ενιαία αγορά δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται μόνο από βιομηχανικούς κανόνες, αλλά θα πρέπει να προβάλλει και κάποια πρότυπα, όπως το διοικό σύστημα. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Ματσόνε ποια είναι η άποψή του, ε, πώς μπορεί να υπάρχει ένα, μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις ανάγκες και αφετέρου στο να ανανεωθούν ε, τα προγράμματα αναδιανεμητικά και άλλα, προγράμματα διανομής και άλλα, ε, μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι μια νέα πρόκληση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τους ε, άλλους ε, συνομιλητές. Έχουμε μπροστά μας ε, την αναγκαιότητα να παντρέψουμε την αναγνώριση της αξίας του δημιουργού ενός έργου μέσα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει κανένας είδους εμπόδιο. Γίνεται τώρα στην Ιταλία λόγος για μια οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να ορίσουμε τους κανόνες όσον αφορά τους service provider χωρίς να αγγίξουμε τον τελικό χρήστη, χωρίς να υπάρξει και το ενδεχόμενο κυρώσεων ή μήπως πιστεύετε ότι η ελεύθερη πρόσβαση που πρέπει να ισχύει για όλους ε, στα προγράμματα του διαδικτύου αυτή θα πρέπει να λάβει μια προληπτική μορφή, δηλαδή συμφωνίες ανάμεσα στους ε, παραγωγούς, όλα εκείνα τα οποία είναι θετικά και ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ισχυρά φαινόμενα ε, πειρατείας. Φαινόμενα τα οποία οδηγούν στο να παίρνει κανείς πολλά και να δίνει πάρα πολύ λίγα Μήπως αυτό θα πρέπει να λάβει και μία άλλη μορφή εφαρμογής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπελέτ, εισηγητής για το ε, διοικό σύστημα. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα όπως και ο κύριος Ματσόνε να μιλήσω για το ψήφισμα και την έκθεση που εγκρίναμε εδώ στο Κοινοβούλιο το περασμένο Νοέμβριο και που είναι πολύ επίκαιρη γιατί εδώ πρόκειται για το μέλλον του διπλού συστήματος. Είναι σημαντικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μας προτύπου, το είπε και η κυρία Τρούπελ. θέλουμε παρά την ενιαία αγορά να διατηρηθεί η ποικιλότητα και να υπάρχει το διπλό σύστημα. Αυτό λοιπόν το διπλό σύστημα το επαναλάβαμε και εμείς ως ιδέα στο ψήφισμά μας δυστυχώς απειλείται. απειλείται από την ισχυρή θέση, την κυρίαρχη θέση που έχουν ορισμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών καθώς και η Apple, η Google και η ανεπίσημη διανομής, όχι ο γραπτός τύπος, όχι η δημόσια διανομή και τα δημόσια κανάλια, αλλά το Google και άλλοι τέτοιοι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι φρονούν οι καλεσμένοι μας γι' αυτό. Ποιες λύσεις θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Και ο Πιότρ μίλησε για άλλα πρότυπα, εναλλακτικά εμπορικά πρότυπα. Ποια είναι αυτά τα εναλλακτικά πρότυπα. Είναι το σύστημα χαντόπι το γαλλικό, ποιο είναι. Όλα αυτά έχουν επικριθεί. Γιατί νομίζω ότι ψάχνουμε, ψάχνουμε, πρέπει να υπάρχουν κάπου κάποια πρότυπα αλλά να μας τα πείτε. Και τέλος, πάλι για εκείνον που εκπροσωπούσε την Νόκια, αυτά που είπε μας ανησύχησαν πολύ. Τα είπε σίκα σίκα σκάφη σκάφη και το ψηφιακό πρόγραμμα που είναι για μας πολύ σημαντικό πρέπει να ξέρουμε αν είναι εφαρμόσιμο. Μήπως άθελά μας στρώνουμε το δρόμο για τις μεγάλες αμερικανικές και ασιατικές επιχειρήσεις απλώς και καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τι να κάνουμε λοιπόν. Αν πραγματοποιηθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά θέλουμε να ξέρουμε αν δεν θα μας πνίξουν αυτές οι μεγάλες ασιατικές και αμερικανικές επιχειρήσεις που θα έρθουν να μας πάρουν το ψωμί από το στόμα. Σουλούς. Ευχαριστώ. Σε όσους ασχολούνται με τον κινηματογράφο θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί η μετάφαση... στα ψηφιακά να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα να μεταφερθούν δηλαδή τα παραδοσιακά κινηματογραφικά έργα στο ψηφιακό υπόβαθρο. Οι δε διαφημιστέ πώς θα περάσουν από, το, από τη μία μορφή στην άλλη. Φαίνεται ότι το φοβούνται. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερες επεξηγήσεις χρειάζονται. Τώρα θα ήθελα να παρακαλώσω τους ε, εμπειρογνώμους να απαντήσουν. Ο κύριος Ματσόνε θα λάβει πρώτος το λόγο, έχει λάβει και τις ε, περισσότερες ερωτήσεις. Να είστε σύντομος παρακαλώ, ή δυνατόν. Πάρα πολλές ερωτήσεις μου ετέθησαν ναι. από τους ε, διάφορους ε, ομιλητές και αγορητές. Να απαντήσω πρώτα στην κυρία Τρούπελ ότι Ε, μιλούσαμε για την ουδετερότητα του δικτύου, για διαφάνεια. Δύσκολη η ερώτηση, αλλά εγώ να σας ξεκαθαρίσω όσο γίνεται. Διαχείριση κυκλοφορίας διάφανη σημαίνει ότι οι πάροχοι του ίντερνετ θα πρέπει να μην κάνουν δυσμενείς διακρίσεις και κοιτάξτε τι είχε με την Comcast. Μέχρι το αποκαλυφθεί, είχαν προβεί σε θερμενεί διακρίσεις. Και όλοι νομίζανε ότι κάτι συμβαίνει με τη σύνδεση. Όχι, δεν ήταν η σύνδεση. Έφταγε η διαχείριση. Έφταγε η διαχείριση που έτσι παραβίαζε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Άρα χρειάζεται να μην πάνε μια κρίση, να ξέρει ο κόσμος Χρειάζονται εγγύησεις και προς την βιομηχανία και προς τον ε, καταναλωτή στο τοπίο. Ιντερνετ υψηλής ταχύτητας. Δεν το είπα ως θεμελιώδες δικαίωμα, σέβομαι την... και συμφώνω με την άποψή σας που το είπατε εσείς. Το θέμα είναι όμως ποιος φέρει το κόστος. Συνήθως αυτό είναι θέμα νομοθέτη. Να σας πω όμως τις ιδέες μου. Υπάρχει εδώ κάτι βασικό. Είναι θέμα φάσματος. Η ζήτηση για το ίντερνετ και κυρίως ε, μέσω κινητού τηλεφώνου, το mobile internet ή κινητή συσκευής συνέχεια αυξάνει, έχουμε αυτή την point to -point communication στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα, ήταν ένα σήμα που πήγαινε σε κάποιον, που επισήμωνα πήγαινε σε όλους, όμως από το, εν, από το ένα σε πολλούς, ε, τώρα έχει γίνει από πολλούς σε πολλούς, άλλαξε το τοπίο. Το δε, βέβαια, φάσμα και αυτό θα είναι σε σπάνιδα εάν όλα τώρα ανοίξουν. Όμως, όσον αφορά το Ιντερνετ υψηλής ταχύτητας, δεν, αυτό είναι θέμα που ξεπερνάει το φάσμα. Χρειάζεται περισσότερο φάσμα, περισσότερη ζήτηση και άρα παραχωρείται κομμάτι του δημόσιου χώρου. Γιατί υπάρχει πολλή ζήτηση. Όμως, είναι σωστό αυτό ή πρέπει ο νομοθέτης να βρει ένα μια άλλη λύση. Ποιε είναι οι προτεραιότητες. Μήπως χρειάζεται το Ιντερνετ υψηλής ταχύτητα κυρίως στην Ήπεθρο ώστε να μην έχουμε αστιφιλία. Να μην έχουμε δυσμενή διάκριση βάρο του. Πολλά θέματα. Εγώ απλώς τα αναφέρω. Ευτυχώ, ευτυχώ δεν έχω τι δικέ σα ευθύνε. Τώρα όσον το ψηφιακό διαβατήριο και το επάγγελμα. Αυτό αφορά κυρίως καταναλωτές. Οι, οι, οι broadcasters οι φορείς τέλο πάντων που αναμεταδίδουν, που παρέχουν ε, θα πρέπει να χειριστούν το θέμα του μέσω ποιας πλατφόρμας θα γίνεται η παροχή, η μετάδοση. Όσο πιο πολλέ ενεργέ έχουμε, τόσο καλύτερα. Κάτι άλλο τώρα, όπω είπε, εδώ είναι η συνάδελφοι που λέμε το, το λόγο, ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται με τα όρφανα έργα, είναι τα, τα έργα που δεν ξέρουμε, Ποιο είναι ο δικαιούχο, ο αποδέκτης, τον ανταμοιβή. Το ίδιο λοιπόν και όσον αφορά την δημόσια πρόσβαση στο ίντερνετ, ναι, θέλουμε να πληρώσουμε, δεν ξέρουμε σε ποιον. Να, παράδειγμα. Δουλεύω στη ΡΑΕ, εντάξει. Η ΡΑΕ, λοιπόν, προσφέρει βίντεο με ψηφιακή τεχνολογία 200.000 ε, έργα, κομμάτια. Πόσα 200.000 από τα 2 εκατομμύρια γιατί. Για τα υπόλοιπα των 2 εκατομμυρίων δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δικαιούχος για τα σχετικά δικαιώματα. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα παρέχουμε και αυτά. Ένα, ας πούμε, μια συναυλία στη σκάλα του Μιλάνου, θυμάμαι, κάναμε ένα τεστ. Μετά 50 χρόνια πρέπει 220 που ήταν, έπρεπε να δούμε αν ζουν, αν έχουν κληρονόμους, αν είναι παντρεμένοι, πόσα παιδιά έχουν, ε, τι γίνεται, έχουν από δεύτερο γάμο άλλα παιδιά κλπ. κλπ. Αυτό για να καταλάβετε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Ο κ. Καβαντά τώρα μας είπε για το πώς θα εξασφαλίσουμε την συνέχεια και συνέχιση και στην ποιότητα της μετάδοσης, της διάδοσης των έργων. Εδώ είναι βασικός ο ρόλος του δημοσίου, περιεχόμενο ποιοτικό, μαθαίνουμε λένε και περισσότερο πώς να ε, δημιουργήσουμε σε διαφορετικές πλατφόρμες αυτή είναι η δουλειά μας βέβαια σε μερικές χώρες δεν, δεν, δεν μας το ζητάνε να το κάνουμε δυστυχώς και αν δείτε την καμπύλη όλα είναι και περισσότεροι προσφεύγουν στο ίντερνετ για οπτικοακουστικά. Και μερικοί, μερικά από τα μέλη μας ε, έχουν υφίσταται δεσμένη διάκριση γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω στο ίντερνετ με το κοινό του. Όσον αφορά το, το περιεχόμενο και τη δεσμενή διάκριση, δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση για μην έχουμε δυσμένη διάκριση στο περιεχόμενο. Όπως ξέρετε, στην Ορβηγία έχει γίνει μια συλλογική σύμβαση με όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι μια λύση. Όσο δουλεύει, δουλεύει. Όμως, θα πρέπει τότε να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο. Το ιδιωτικά αντίγραφα. Νομίζω οι συνάδελφοι το ανέφεραν, αυτοί μπορούν να αποφασίσουν, αλλά βέβαια. Τι. I stop now and I come back with Miss Costa. Because they said me that I have to be afraid of, of you because you said... Τι να σου πω, έχω δύο αγόρια και καταλαβαίνετε, τα ξέρω. Τι είναι, εννοεί ότι... <laughs> Η κυρία Πάκ εκτός μικροφώνου. Πάκ. Ματσόν. Πάμε τώρα στο πρόβλημα των πόρων. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, δεν σας έδειξα προηγουμένως τις διαφάνειες γιατί δεν υπήρχε χρόνος, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος από την Νόκια, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, κανονισμούς ε, που καλύπτουν ε, ένα κομμάτι των διαθέσιμων πόρων. Όσα εκείνους δηλαδή που περνούν ε, μέσα από το κύκλωμα του broadcasting και του κινηματογράφου. Και αυτή τη στιγμή κονδύλια μεταφέρονται από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο προς το διαδίκτυο. Η, αυτά όσον αφορά τη γραμμική κατανάλωση, τη μη γραμμική κατανάλωση, εκεί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές δυνάμεις στην αγορά. Η γραμμική κατανάλωση στην Ευρώπη είναι ακόμα πολύ μεγάλη στην Ευρώπη. Οι δικοί μας οι broadcasters κυριαρχούν ε, στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε όμως για το video on demand, εκεί ε, αλλάζει τελείως, ο συσχετισμός των δυνάμεων όσο περισσότερο γίνεται κατανάλωση της τηλεόρασης, τόσο περισσότερο μετατίθενται οι πόροι, κυρίως ε, της ε, διαφήμισης. Είπα προηγουμένως, ε, αναφέρθηκα στην Google, στην Apple και σε άλλους που δεν καλύπτονται από κανόνες, δεν υπάγονται σε κανονισμούς. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στη Γαλλία όταν προέκυψε η κρίση του κινηματογράφου τη δεκαετία του 70 η η γαλλική κυβέρνηση είπε ότι γι' αυτό φταίει η τηλεόραση και είπε να πλώσει η τηλεόραση και τον κινηματογράφο γιατί ο κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι της ε, πολιτιστικής μας ταυτότητας. Τώρα, τι γίνεται σήμερα. Εγώ το θέμα ε, το βλέπω προσωπικά αλλά μπορείτε κι εσείς να πείτε τη δική σας άποψη. Το τελευταίο ερώτημα νομίζω το υπέβαλε ο κύριος Μπελέτ. Ε, αυτό θα πω και μετά κλείνω, σας το υπόσχομαι δεν ξαναμιλήσω. Ο κύριος Μπελέτ αναφέρθηκε στο θέμα του τύπου. Ε, για μας ε, ο τύπος, ο τύπος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς, το ομολογώ αυτό, αλλά και πάλι δεν είναι ότι ε, δεν υπάρχουν προγράμματα, παράγονται προγράμματα στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι τα προγράμματα αυτά είναι δωρεάν και κανείς δεν πληρώνει για αυτά. Και κατόπιν Υπάρχει και ένα θέμα που με φοβίζει πάρα πολύ. Πρόκειται για τον αριθμό ε, των πηγών που υπάρχουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ε, του Πανεπιστημίου ε, του Κέμπριτζ για τις πηγές ενημέρωσης που υπάρχουν. Περιορίζονται αυτές οι πηγές όσο ε, λιγότερους ξένους ανταποκριτές ε, στέλνει κανείς στο εξωτερικό, ε, τόσο λιγότερες πηγές ενημέρωσης υπάρχουν. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη ενημέρωση στο διαδίκτυο. Αν όμως δείτε προσεκτικά θα δείτε ότι είναι τέτοια πράγματα που επαναλαμβάνονται από λιγότερες πηγές. Αυτό φοβίζει, ναι με φοβίζει εμένα ως πολίτη, όχι ως EBU αλλά ως πολίτη με φοβίζει αυτό. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήμουν τόσο αυστηρή γιατί οι περισσότερες ε, ερωτήσεις απευθύνθηκαν σε εσά ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Νόκια. Ε, θα ήθελα να είμαι πολύ σύντομος, αλλά εγώ θα απαντήσω ε, στο θέμα της ευρυζωνικής ε, πρόσβασης και ποιος ε, πληρώνει. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ περίεργη. Ένα κομμάτι πληρώνεται από τις διαφημίσεις και κατόπιν υπάρχει ένας τομέας που χρειάζεται την δημόσια υποστήριξη. Δεν λέω βέβαια ότι όλες οι χώρες και όλες οι περιοχές πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ καλά μοντέλα στην Ευρώπη. Εγώ έρχομαι από την Φινλανδία, ε, έχουμε υποσχεθεί ε, μεγάλη διάδοση της ευρυζωνικότητας σε όλα τα νοικοκυριά σε μια ε, χώρα με μεγάλες αποστάσεις και χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε χρήματα για να καλύψουμε τη ζήτηση μιλάμε για κονδύλια του Ταμείου Συνοχής και κονδύλια που συγκεντρώθηκαν από, τις, από τη χορήγηση αδειών. Υπάρχει λοιπόν δημόσια δέσμευση και χρηματοδότηση και αυτή είναι μια απόφαση που λάβαμε. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχουν χρήματα, ε, το θέμα είναι απλά και μόνο να ληφθούν οι απαραίτητες ε, αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στις ερωτήσεις ε, που μου ετέθησαν, θέλω να πω το εξής, θα τα απαντήσω όλα μαζί. Ε, όσον αφορά τα ιδιωτικά αντίγραφα, όταν έχουμε ένα CD Μπορούμε να το παίξουμε στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο, στο σκάφος μας. Τώρα, αν κάνουμε ψηφιακό αντίγραφο, πρέπει να πληρώσουμε τέσσερι φορές και κάθε φορά πρόκειται για ιδιωτικό αντίγραφο ή όχι. Αυτό δεν είναι σαφές ούτε για τον καταναλωτή, ούτε για τον ε, φορέα παροχή ούτε για κανέναν. Δεν υπάρχει ορισμός του τι είναι ιδιωτικό αντίγραφο. Μερικοί λένε όταν χορηγείται άδεια ε, σε ένα πρόγραμμα, δεν χορηγείται άδεια και για ιδιωτικό αντίγραφο. Και πάλι αυτή είναι μια τελείω διαφορετική ερμηνεία σε διάφορα μέρη τη Ευρώπη σε ορισμένα μέρη, σε ορισμένες χώρες κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, σε άλλες πάλι όχι. Έχουμε διαφορετικούς ορισμούς για το ιδιωτικό αντίγραφο και πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση ε, ως προς τον ορισμό. Κατόπιν, σωστή αποζημίωση. Η οδηγία λέει ότι η αποζημίωση πρέπει να βασίζεται ε, και στην πραγματική ζημιά, ε, να βασίζεται στην σωστή και δίκαιη αποζημίωση. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να έχει σχέση και με τη μνήμη του PC. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μνήμη αυτή για τα email, για τις φωτογραφίες, για δικά μας προγράμματα. Ε, εδώ η αποζημίωση δεν είναι δίκαιη. Πρέπει να ορίσουμε τι είναι δίκαιη αποζημίωση και να υπάρχει και ένα μέτρο του πώς μετράμε αυτή την αποζημίωση. Ε, κατά κανόνα δεν έχουμε ανεξάρτητες έρευνες στα κράτη-μέλη για να δούμε ε, ποιο τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για τα ιδιωτικά αντίγραφα. Και τρίτον, αμοιβέ. Εμείς ε, τα σώμεθα ανεπιφύλακτα υπέρ του ότι ο καλλιτέχνης και όποιο έχει τα ε, δικαιώματα copyright πρέπει να αμείβεται. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη αρχή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να γίνει κάτι τέτοιο ως έχει το σύστημα σήμερα. Δεν βλέπουμε να αμείβεται σωστά ο καλλιτέχνης λόγω του ότι είναι περίπλοκο το σύστημα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά θαυμάσιων εταιριών στην Ευρώπη ξεκινώντας από τη Spotify και άλλες ε, που έχουν φτιάξει ένα σύστημα όπου κάθε κομμάτι μουσικής που κατεβαίνει καταγράφεται και από κάθε κατέβασμα ένα κομμάτι χρημάτων ε, μεταφέρεται στον καλλιτέχνη και ένα τμήμα των χρημάτων μεταφέρεται στην εταιρεία που ε, μαζεύει χρήματα από τις ε, αδειοδοτήσεις. Έχουμε λοιπόν την απαραίτητη τεχνολογία, αλλά το σύστημα που ισχύει εμποδίζει αυτά τα συστήματα να εφαρμοστούν στην Ευρώπη. Έχουμε ένα τέτοιο νομικό σύστημα που αναγκάζει τους ε, καλλιτέχνες να είναι μέλη της, των εταιριών που συγκεντρώνουν τα χρήματα. Και βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους καλλιτέχνες να προσπαθούν να πλοηγήσουν έξω από το σύστημα να συνάπτουν συμβάσεις ε, με τους ε, φορείς ε, του διαδικτύου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο, το εμπόδιο είναι εκείνο που μας εμποδίζει σήμερα ε, να συγκεντρώνουμε χρήματα από το διαδίκτυο. Και αυτό λόγο υποφέρουμε από την πειρατεία. Διότι η πειρατεία είναι το αποτέλεσμα του ότι δεν υπάρχει ένα ικανοποιητικό σύστημα από νόμιμες αναγνωρισμένες πηγές. Και γι' αυτό υποφέρουμε από την πειρατεία. Και τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Ολλανδία. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, την αγορά θα την αφήσουμε θα την εγκαταλείψουμε στους Αμερικανούς παίκτες. Αν όμως είχαμε μια νέα αγορά, τότε εταιρείε όπως η Spotify και άλλες ε, θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερης κλίμακας, να υπηρετήσουν τους ε, Ευρωπαίους ε, καταναλωτές, να προβάλλουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εκτός Ευρώπης. Μπορεί κανείς να είναι ε, αντίπαλος της Google και άλλων, αλλά όσο δεν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα, εμείς ε, απλά και μόνο ε, θα κάνουμε τη διανομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Σουάρες Λουτσάνο, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Pardon τι είπατε, Το περισσότερο τα είπαμε παρακαλώ μόνο πέντε λεπτά γιατί έχουμε και άλλα και άλλους να ακούσουμε. Is... Πρώτη μου ερώτηση, το Αθάνο. Είπαμε λοιπόν, για δημιουργούς, για, ερ... για ερμηνευτές. Δεν έχουμε πει για τους παραγωγούς όμως. Γιατί ο παραγωγός είναι στη δημιουργική βιομηχανία το κλειδί. Όπω είπε το κρατικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκού Διοκτησία έχει την πρωτοβουλία και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα όσα γίνονται ή στην παραγωγή. Δηλαδή αναλαμβάνει το κίνδυνο, το ρίσκο. Χωρίς παραγωγό δεν υπάρχει οπτικοακουστικό. Δεύτερο θέμα, δεύτερη ερώτηση. Εάν η αγορά είναι ανοιχτή και διαθέσιμη, γιατί τότε οι Αμερικάνοι δεν είναι ήδη στην παραγωγη δηλαδη αναλαμβανει το κινδυνο το ρισκο χωρι παραγωγο δεν υπαρχει οπτικοακουστικο δευτερο θεμα δευτερη ερωτηση εαν η αγορα ειναι ανοιχτη και διαθεσιμη γιατι τοτε οι αμερικανοι δεν ειναι ηδη στην αγορα και αυτό θα πρέπει να το αναρωτηθούμε. Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Βρετανική αγορά. Τι έγινε. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την προσφορά. Και όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, ελπίζουμε θα έχουμε και την ουδετερότητα. Στους Financial Times πριν από δύο χρόνια η Μακέζη Κολσάντ έλεγε ότι 300 δις ευρώ είναι αυτά τα οποία απαιτούνται για την αγορά. Αλλά ποιος θα το πληρώσει, οι καταναλωτές να επιδοτήσουν τις ε, επιχειρήσεις. Επίσης μιλάμε για αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Ήδη έχει αλλάξει. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε την προσαρμογή του μοντέλου. Είναι θέμα επιβίωσης. Αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ σαφές. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται και πληρώνουν την ύφη η παραγωγή, οι ερμηνευτές. Αυτοί το στηρίζουν και δεν έχουν αποζημιωθεί. Το γίνεται τώρα με το δυτικό αντίγραφο. Το περισσότερο θέμα για το δυτικό αντίγραφο τα έχει κρίνει ε, μέχρι και την, ε, τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην αρχή μια απόφαση το ορίζει και λέει ότι είναι αντίγραφο για προσωπική χρήση του αντιγραφέα. Θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν μιλάμε εδώ τώρα για την έννοια. Μιλάμε για την ποσότητα. Το κάθε αντίγραφο που φτιάχνεται από αυτόν τον τρόπο είναι ξεχωριστό ιδιωτικό αντίγραφο. Τα όρια βέβαια είναι σαφή και λύσει την απόφαση ότι θα πρέπει να πληρωθεί. Από τον καταναλωτή που θα το χρησιμοποιήσει με τα μηχανήματα που έχει. Και επίσης λέει το κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει την ε, αποζημίωση στις εταιρείες εκείνες που έφτιαξαν το δημιούργημα το οποίο, το οποίο κάποιος γι' αυτό και πριν το iCloud η Apple πλήρωνε μεταξύ 100 και 150.000 δολάρια στις ε, εταιρείε δίσκων. Είναι τα όρια του ιδιωτικού αντιγράφου. Thank you very much. Now... Πακ, ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Παρό τώρα όσον αφορά τον κινηματογράφο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η ψηφιακή μετάβαση και η το, το, το, το, του που θα καταλήξουν όλα αυτά μας έχουν να πούμε ότι σήμερα έχει σχεδόν γίνει εν μέρει όσον αφορά την εκμετάλλευση στην Ευρώπη. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες και σε, αυτές, σε αυτούς τους κινηματογράφους δίνουμε μόνο ψηφιακά έργα. Τώρα οι μεγάλη και οι ανεξάρτητοι δεν υπάρχει Ευρώπη δύο ταχυτητών. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Όλοι θέλουν να είναι ψηφιακοί. Και σας τονίζω ότι εάν υπάρχουν κάποιες ζημίες, εάν κάποιοι μετογράφοι πρέπει να κλείσουν, εάν πρέπει να κλείσει κάποια εταιρεία διανομής, τότε σας επισημαίνω ότι αυτό δεν θα είναι ε, κάτι που θα χτυπήσει τις, ε, τις κινηματογράφους multiplex είτε τους μεγάλους της διανομής. Θα είναι οι ανεξάρτητοι που θα κλείσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκεί θα είναι οι ζημίες. Και βέβαια ξέρετε ότι όταν κοιτάτε τι προγράμματα παίζει ο κινηματογράφος στην Ευρώπη, εθνικός κινηματογράφος, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος εκπροσωπείται λιγότερο στα multiplex παρά στους ε, ανεξάρτητους. Το, το, το, το, το, μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσπάθειας το εξασφαλίζουν οι ανεξάρτητοι για τα ευρωπαϊκά έργα. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις ούτως ώστε η μετάβαση να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορη αλλά για τους διανομείς και για τους κινηματογραφιστές τους ανεξαρτήτους. Κύριε Πάκ, χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πάκ, συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο. Η κυρία Αλεξάνδρα Περτσκαλίνσκα, εξ ονόματος της Πολωνικής Παροεδρίας. Πρέπει και εσείς να σεβαστείτε όμως τον ίδιο χρόνο ομιλίας. Ορίστε κυρία Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και διότι μας επιτρέπεται να λάβουμε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και τους εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σχεδιαγραφήσω έτσι τηλεγραφικά τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για τα οπατικοακουσιτικά. Πρώτον, η ψηφιοποίηση των περιεχομένων και ιδιαίτερα της κληρονομιάς στο, του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών είναι κάτι που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες δεν διευκολύνουν μόνο τη διατήρηση παλαιών έργων αλλά επίσης τα καθιστούν πιο προσβάσιμα στον ευρωπαϊκό λαό και στο ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό βέβαια έχει θέσει και νέα ερωτήματα ως προς το ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών που δίνουν πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά και τη διατηρούν. Επίσης το Ευρωπιάνα, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι σημαντική για μας γιατί θεωρούμε ότι ο ρόλος του, της στη νέα ψηφιακή σκηνή θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Χρειάζεται λοιπόν η κατάλληλη χρηματοδότηση. Γι' αυτό η Πολωνική Προεδρία προτείνει την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διατήρηση των οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών έργων και τα θέματα του copyright ή των δικαιωμάτων όπως συζήτησαν οι υπουργοί στην άτυπη συνεδρίασή τους στο Βρότσλαφ θα συζητήσουν στις 9 Σεπτεμβρίου. Επίσης θέλω να τονίσω το θέμα της ασφάλειας προστασίας των ανηλίκων. Ξέρουμε ότι η ψηφιακή εποχή άλλαξε πολλά πράγματα και τα παιδιά και οι νέοι είναι οι πιο μεγάλοι γνώστες της. Απ' την άλλη είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα γιατί δεν γνωρίζουν πάντοτε τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν από το video on demand. Γι' αυτό θα θέλαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στο Συμβούλιο για την προστασία των ανηλίκων. Στα πλαίσια ίσως της δέσμης προτάσεων για το ασφαλέστερο ίντερνετ. Τώρα για την κυκλοφορία και διάδοση των οπτικοακουστικών έργων στην Ευρώπη είναι επίσης σημαντικό νομίζουμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Media ε, θα εγκρίνουμε μάλλον την επόμενη προγραμματική περίοδο γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι η δημιουργία στον οπτικοακουστικό και ιδιαίτερα κινηματογραφικό τομέα είναι το κυριότερο θέμα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα Μίδια θα ανταποκρίνεται στους στόχους του ως προς την ψηφιοποίηση κινηματογραφικών έργων. Επίσης πολύ σημαντικό, επίσης και θα θέλαμε να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός κινηματογράφος θα είναι μια ευκαιρία που δεν θα τη χάσουμε γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στην Ένωση να εξοπλιστεί με τα εργαλεία που χρειάζεται για να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνοχή και σε αυτό το θέμα. Αυτό οικονομικά βέβαια σημαίνει ε, ισχυρή χρηματοδότηση και θεωρούμε ότι μια βιώσιμη χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν η Ένωση τη χορηγήσει. Γιατί πρόκειται για ένα μοναδικό σχέδιο πολυπολιτισμικό. Δεν μπορεί βέβαια να υπάρξει μία ενιαία ομοιόμορφη δημόσια ενίσχυση θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον, θα ζητήσουμε χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά όπως θα χρειάζεται αναπερίπτωση. Και τώρα με την άδειά σας θα δώσω το λόγο στον ε, πυρογνώμονά μας για τα πνευματικά δικαιώματα, ο κύριος Ομπάνσκι. Ομπάνσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με την άδειά σας ε, θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Το copyright έχει αναφερθεί στη συζήτηση ως θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την ψηφιοποίηση και την πανευρωπαϊκή διάδοση των έργων. Η νομοθεσία των πνευματικών δικαιωμάτων όμως δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως φραγμός ως προς την πρόσβαση σε περιεχόμενο και στη δημιουργία της έννοια ψηφιακής αγοράς αλλά ως πρόσθετο κίνητρο για τους δημιουργούς και πιστεύουμε ότι η βιομηχανία αυτή πρέπει να επωφεληθεί και αυτή από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα περιεχόμενα με όλους τους δυνατούς νόμι, νόμιμους τρόπους. Επίσης πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των έργων που δεν μπορούν, δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν όπως ε, έργα εκτός εμπορίου ή έργα χωρίς συγγραφέα. Πρέπει να λυθούν αυτά τα διάφορα νομικά προβλήματα για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Στο ψηφιακό πρόγραμμα για την Ευρώπη τα προβλήματα αυτά έχουν αναφερθεί και πιο πρόσφατα ακόμα στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την ενιαία αγορά για ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης για την πρόσβαση αυτή η Κομισιόν πρότεινε να ταυτιστούν και να διατεθούν και τα έργα χωρίς συγγραφέα. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες της Προεδρίας μας και θα προσπαθήσουμε να τα πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήδη στην ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο αρχίσαμε να τα συζητούμε, αλλά βέβαια το θέμα είναι μεν σημαντικό, αλλά είναι απλώ ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Αγορά που δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα που αφορούν τη διαμεθοριακή ε, διάδοση, παγκόσμια μάλλον, διεθνή διάδοση όλων των έργων. Έχει γίνει μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό που δημοσιεύτηκε μόλις σήμερα. Τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν. Και πρόκειται η Κομισιόν να κάνει και πρόσθετες προτάσεις σε λίγο. Αυτές οι πρόσθετες πρωτοβουλίες νομίζουμε θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στα έργα ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν ότι θα διατηρείται με ίσους όρους η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της Ευρώπης ε, χωρίς να παραβιάζονται και τα πνευματικά δικαιώματα και τα έσοδα των δημιουργών. Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας μας είπα και πριν ότι θα τονίσει ιδιαίτερα τα έργα χωρίς συγγραφέα και αν η πρόταση για τη συλλογική διαχείριση τους γίνει δεκτή φέτος θα το προωθήσουμε δεόντως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Και το περιεχόμενο, ε, και το περιεχόμενο. Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο για το ίδιο θέμα στην Κομισιόν, την οποία ευχαριστώ για την παρουσία της. Ο κύριος Ντρέτεν Μπράι, παρακαλώ. Που αν δεν απατώμε είναι Γερμανός, από τη Γενική Διεύθυνση Πληρόφ. Ε, Αυστριακό είναι το όνομά μου. Είναι η κοινή γλώσσα που μας χωρίζει. Σήμερα θα είμαι πολύ σύντομος ε, γιατί έχουμε και άλλους εμπειρογνώμονες ε, από άλλους τομείς που θέλουν να ασχοληθούν με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ε, θέματα. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ευριακή τηλεόραση και την Connected TV. Ο κύριος Ματσόν κατά κάποιον τρόπο είπε ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες τώρα που έχουμε το διαδίκτυο ε, στο διαδίκτυο τηλεόραση. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι το ίδιο μέσο, είναι ένα, μια συσκευή. Μια συσκευή που ε, προσφέρει ε, μη γραμμικές υπηρεσίε και έχουμε την τηλεόραση που προσφέρει γραμμικές υπηρεσίες. Από την άλλη, οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οι ανανέωση ή ο της ε, οδηγίας για την τηλεόραση θίγει αυτά τα θέματα. Τα κριτήρια τα ποιοτικά είναι ίδια και για τις γραμμικές και για τις μη γραμμικές ε, υπηρεσίες. Ε. Οι κανόνες για, για ομιλίες που υποδαβλίζουν το μίσος είναι οι ίδιες ή για την προστασία των νέων. Είναι οι ίδιοι οι κανόνες. Η βασική διαφορά αφορά στις, ε, στους ποσοτικούς ε, κανόνες ε, διαφήμισης και αυτό συζητιέται διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα με, τα, με τη διάρκεια σε λεπτά για την κρατική τηλεόραση, αλλά για την ε, ιδιωτική τηλεόραση τίθεται το θέμα της περαιτέρω φιλελευθεροποίησης ε, για γραμμικές υπηρεσίες για την ε, τηλεόραση. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις προδιαγραφές. Εκεί υπάρχουν δύο θέματα που ετέθησαν σήμερα τέθη το ερώτημα αυτό δεν αποτελεί ε, πρόβλημα για τους παραγωγούς. Αυτό δεν εμφανίστηκε μέχρι τώρα στις συζητήσεις μας γιατί το διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό έχει τυποποιηθεί. Εκείνο που συζητήθηκε είναι ένα θέμα που αφορά ε, το σημείο επαφής με το χρήστη. Ε, εκεί λοιπόν ένα κανάλι που εκπέμπει στο Βέλγιο έχει διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικούς ε, χρήστες που ε, ανακαλούν διαφορετικά προγράμματα από κάποιον που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γερμανία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομος ε, και αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αφορούν την ψηφιακή αγορά, την κοινή αγορά Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί ε, εγκρίνεται, θα θεσπιστεί η πράσινη ε, βίβλος και η συναδελφός μου είναι αρμόδια και έχει ε, το λόγο. Πράγματι, έχετε το λόγο γιατί σήμερα εγκρίθηκε η πράσινη βίβλος και ίσως μπορείτε να μας θέσετε και τις λύσεις και όχι μόνο τα ερωτήματα. Η δική μου η παρέμβαση θα είναι πολύ σύντομη αφορά κυρίως τις ερωτήσεις. Πρόκειται για ένα πολύ ε, εκτεταμένο και περίπλοκο θέμα. Πολλοί έθιξαν διάφορα ερωτήματα. Εμείς ξεκινάμε με ορισμένα βασικά. Καταρχήν, η ε, πολιτιστικές ε, βιομηχανίες είναι πολύ σημαντικές ε, στην Ευρώπη, όχι μόνο οικονομικά αλλά και για κοινωνικούς λόγους. Έχουμε τις οπτικοακουστικές αγορές που μέχρι τώρα ήταν εθνικές για όλους αυτούς τους λόγους που ετέθησαν σήμερα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παράγει και οι διανομείς έχουν πλέον το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο παρέχουν στους καταναλωτές και είναι και διαφορετικός ο τρόπος πρόσβασης ε, στο υλικό αυτό και έρχεται ένα σημαντικό ερώτημα το κατά πόσον οι ρυθμιστικοί φραγμή ε, στην Ευρώπη παρεμποδίζουν ε, νέες παραγωγές, νέα πρόσβαση και κατά πόσον προσφέρουν σωστή αποζημίωση ε, στους καλλιτέχνες ε, και στους ε, συγγραφείς. Στην Πράσινη Βίβλο παρουσιάζουμε την κατάσταση και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι ο οπτικοακουστικός τομέας είναι τελείως διαφορετικός από, το, από τη μουσική. Στον τομέα της μουσικής ε, έχουν ε, γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για συλλογικές αδειοδιοτήσεις αλλά όπως ακούσαμε στον οπτικοακουστικό τομέα εξετάζουμε κυρίως την κατάσταση ε, μεμονωμένων αδειών. Οι παραγωγή ταινιών κατά κανόνα έχουν όλες τις στα χέρια τους και το πλαίσιο του copyright δεν παρεμποδίζει πανευρωπαϊκές αδειοδοτήσεις οπτικοακουστικού υλικού. Ίσως να υπάρχουν οικονομικοί φραγμοί και γι' αυτό κατά κύριο λόγο έχουμε εθνικές αγορές όπου οι παραγωγοί πουλάνε ε, πάνω σε εδαφική βάση. Εξάλλου υπάρχουν και πολλές σημαντικές ε, γλωσσικές διαφορές όπου το οπτικοακουστικό υλικό ε, δεν είναι τόσο διασυνοριακό όπως η μουσική γιατί υπάρχει το θέμα του υποτιτλισμού, του μεταγλωτισμού ε, πόσο μάλλον και θέματα ε, ε, γούστου προσέγγισης. Το θέμα είναι ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα για τον οπτικοακουστικό τομέα. Ποια είναι η κλίμακα και το εύρος. Και αυτά τα εξετάζουμε σε σχέση με την αναμετάδοση πέρα από τα σύνορα, τη μετάδοση, video on demand, και επίσης ε, και σε σχέση με τις ε, ευρωπαϊκές παραγωγές γνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή ε, διέπεται από διαφορετικά κριτήρια. Οι παραγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατακαιρματισμένοι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς στη γενική μας τη διεύθυνση το, παίρνουμε ιδιαίτερα, το λαμβάνουμε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη μας. Ως εκ τούτου τους άμεσα ενδιαφερόμενους τους καλούμε να μας πούνε ποια είναι η κλίμακα και το μέγεθος του προβλήματος. Τους καλούμε να λάβουν υπόψη τους σε διάφορες αναλλακτικές λύσεις ανάλογα με το πρόβλημα και αυτές ξεκινούν από το πλαίσιο συλλογικών αδειοδοτήσεων ε, στο οποίο είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι. Ε, θέτουμε επίσης ε, ερωτήματα σχετικά με έναν εναρμονισμένο κώδικα copyright Επίσης ε, θέτουμε ερωτήματα για τη χρήση της, για την αρχή της, ε, για τη χρήση της αρχής ε, προέλευσης. Αυτά είναι ερωτήματα με πάρα πολλές προεκτάσεις. Στο δεύτερο σκέλος ε, της Πράσινης Βίβλου ασχολούμεθα με την αποζημίωση ε, των ε, δημιουργών και των καλλιτεχνών και είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό όσοι δημιουργούν να αμείβονται σωστά. Και λέμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και κατόπιν ε, θέτουμε το ερώτημα της σωστής χρήσης οπτικοακουστικού υλικού που σημαίνει και πρόσβαση από άτομα με αναπηρία. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν εδώ και τέλος ε, θέτουμε ένα ερώτημα σχετικά με τις ειδικέ ανάγκες ε, ε, θεσμών πολιτιστικής κληρονομιάς, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ινστιτούτα αυτά στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για μελλοντική χρήση. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω και για άλλα θέματα copyright αν θέλετε ή αν θέλετε μπορώ να σταματήσω εδώ γιατί αυτά αφορούν στην πράσινη βίβλο για τα οπτικοακουστικά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντόλμπι, λέει η Πρόεδρος. Ε, νομίζω θα διαβάσουμε την πράσινη βίβλο ε, θα εγερθούν και άλλα επιπρόσθετα ερωτήματα πέρα από αυτά που θέσαμε σήμερα μόνοι μας και που ίσως ε, τεθούν και από τους ε, εμπειρογνώμονες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πολλές απαντήσεις και οι απαντήσεις που δίνουν οι μεν δεν ε, γίνονται αποδεκτές από τους δε. Όσον αφορά το copyright υπάρχουν τόσες πολλές απαντήσεις. Οι απαντήσεις στο θέμα του copyright είναι κατ' ουσίαν ο τετραγωνισμός του κύκλου. Ελπίζω λοιπόν σε αυτό τον τομέα ε, να μπορέσουμε ε, τουλάχιστον να έχουμε μια πλειοψηφική άποψη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες ακούσαμε πάρα πολλά τα οποία ίσως ε, να γνωρίζαμε, ενδεχομένως όχι με τόσες πολλές λεπτομέρειες. Ε, στον εκπρόσωπο του Eurocinema θέλω να του πω ότι βεβαίως ε, συμφωνούμε μαζί σας ότι το πρόγραμμα Media πρέπει να αναλάβει αυτό που θίξατε, δηλαδή να μεριμνήσει να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση μικρών κινηματογράφων. Λέτε είναι μικρή κινηματογράφη. Ε, κοιτάξτε, δεν έχουμε και πάρα πολλά χρήματα και γνωρίζουμε ότι ο κοινό αγώνας μας ε, βοήθησε και εδώ θα συμφωνήσει και η Κομισιόν, ε, στο να υπάρχει το πρόγραμμα Μέντια και να ε, χρηματοδοτείται. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό θα μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι μέχρι σήμερα. Όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα του copyright και άλλα, Όλα αυτά είναι τόσο δύσκολα που πρέπει σε όλους αυτούς τους τομείς ε, ε, να τα εξετάσουμε σε βάθος, κυρίως εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι κατά κύριο λόγο το περιεχόμενο. Γιατί χωρίς το περιεχόμενο μπορεί κανείς ε, ε, να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για το ότι είχαμε αυτή την ευκαιρία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, κατά τους επόμενους μήνες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και ίσως τελικά να φτάσουμε σε αίσιο Εν πάση περιπτώσει, εμείς ε, θα ξαναζητήσουμε τη συμβουλή σας, είμαι σίγουρη και ελπίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ε, θητείας θα βρούμε κάποιες ε, καλές λύσεις. Δεν θα ικανοποιηθούν όλοι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε όλοι από κοινού. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας ε, βασιζόμαστε σε εσά για τους επόμενους ε, έξι μήνες ε, και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την ακρόση και να προχωρήσουμε με το θέμα την εισήγηση του κυρίου Μπόρις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης ο συνάδελφος κύριος Μπόρις, Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος ε, στην ψηφιακή εποχή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω ότι η έκθεσή μου που ετοιμάζω μαζί με τους κοιόδης από διάφορες πολιτικές ομάδες είναι έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο που δεν αφορά μόνο ιδιοκτήτες αιθουσών αλλά και παραγωγούς και δημιουργούς και ηθοποιούς και διανομής οι οποίοι αναμένουν ανυπόμονα την έκθεση αυτή αναμένουν και είπαμε και πριν ότι ζούμε μία ψηφιακή επανάσταση στην Ευρώπη που αποτελεί τεράστια ευκαιρία αλλά όπως όλες οι άλλες επαναστάσεις υπάρχει και μια απειλή για ζημίες και θύματα. Όσοι δεν προστατευθούν από την νομοθεσία θα χαθούν. Εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε κάτι τέτοιο γιατί είμαστε ταγμένοι υπέρ του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου σύνθεση πολλών ειδών τέχνης, χώρο, μουσική και άλλα. Θέατρο. Ο Βιμ Βέντερς είπε ότι δεν υπάρχει καλύτερο εργαλείο από τον κινηματογράφο που να μεταφράζει, να δείχνει καλύτερα την ευρωπαϊκή ψυχή για τις επόμενες γενιές. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στον κινηματογράφο και αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτή την καμπή. Αν καταφέρουμε να τον προωθήσουμε θα αναπτυχθεί πολύ γρήγορα Μερικοί φυσικά πρέπει να βοηθηθούν γιατί δεν έχουν τους πόρους για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή. Στην έκθεσή μας αυτήν λοιπόν υποστηρίζουμε απλώς τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο ο οποίος μεταφέρει πολλές και τεράστιες αξίες. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προώθησης του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της πολιτισμικότητάς του, των γλωσσών του από το σινεμά. Αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τους φραγμούς αυτούς, τότε μετά από τα 100 χρόνια ύπαρξης του παραδοσιακού κινηματογράφου θα προωθήσουμε τον ψηφιακό κινηματογράφο για 500 εκατομμύρια δυνητικούς χρήστες του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα για να γίνει αυτή η πολιτική μετάβαση γιατί όπως είπα είναι μια τεράστια ευκαιρία. Επίσης πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος όπως είπε ο Σίγμουντ Μπάουμαν που θα είναι ο κύριος ομιλητής στην ευρωπαϊκή διάσκεψη, πολιτιστική διάσκεψη έχει πει στο παρελθόν ότι το ευρωπαϊκό σινεμά έχει ως κύριο στόχο του την αλλαγή της αντιμετώπισης της νεολαίας. Το ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, βέβαια πρέπει, στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο πρέπει να αντιτάξουμε την πολύ ρηχή πολιτιστική παραγωγή που μας περιτριγυρίζει. Πρέπει να εκτιμήσουμε δεόντως την αξία που έχει το σινεμά αυτό για τις μελλοντικές γενιές. αξία η οποία δεν είναι προφανής οικονομικά αλλά είναι ικανή να διαμορφώσει αντιλήψεις και να βελτιώσει αλληλοκατανόηση ιδίω σε εποχές κρίσης. Οπότε και δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν ορισμένα ακραία ιδεώδη. Το σινεμά λοιπόν και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι πολύ σημαντικά. Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα λοιπόν. Σήμερα όπως είπαν και οι κύριοι Πουαρό και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν η αγορά για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο είναι πελώρια, τεράστια, κολοσιαία. Πάνω από 100.000 έργα ε, δημιουργούνται κάθε χρόνο στην Ένωση ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείες 700. Υπάρχουν όμως χίλια μάλλον προς 700 και μόνο το 27% δυστυχώς παρόλα αυτά των θεατών βλέπουν τα ευρωπαϊκά έργα. Τα υπόλοιπα έργα που βλέπονται είναι κυρίως αμερικανικά. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, πώς γίνεται αυτό, μήπως γιατί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι λιγότερο ελκυστικός, μήπως έχουν λιγότερη αξία. Κατ' εμένα η ψηφιοποίηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους, για τους παραγωγούς που με το παλιό σύστημα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό κοινό γιατί οι παλιές κόπιες λόγω του υψηλού κόστους των δεν μπορούν εύκολα να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες και άρα δεν είναι προσβατές σε όλους και γι' αυτό τόσο πολλά έργα χάνονται σε αυτήν την κοινή αγορά. Ας φανταστούμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία, ας πούμε, αν ένα έργο αξίζει τον κόπο, σε μια ώρα να μπορεί να φτάσει σε όλους όσους θέλουν να το δούνε στην εθνική τους γλώσσα ή σε μεταφράσεις ε, μεταφρασμένη ήδη στην εθνική τους γλώσσα και έτσι να είναι πρόσβατο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα δεν γίνεται. Άλλο πρόβλημα η σε μεταφρασεις ε ηδη στην εθνικη τους γλωσσα και ετσι να ειναι προσβατο σε ολοκληρη την ευρωπη σημερα δεν γινεται αλλο προβλημα η προσβαση Δυστυχώς, δυστυχώς λέγω, η Ευρώπη έχει ακόμα ένα αόρατο σιδηρούν αραπέτασμα. 16.000 άνθρωποι αναοθώνει στη Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική 40.000. Υπάρχει λοιπόν μια διπλή απειλή εδώ. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τα, οι κινηματογραφικές αίθουσες είναι μικρές με μία ή δύο οθόνες και είναι και πολύ απομακρυσμένες η μία από την άλλη ενώ στη Δυτική Ευρώπη η ψηφιοποίηση έγινε από τα λεγόμενα multiplex από αίθουσες με 9-10 οθόνες και γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια πρόκληση μπορούμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη, συνοχή και η ισότιμη πρόσβαση για, στους Ευρωπαίους πολίτες, για τους Ευρωπαίους πολίτες στο σινεμά και στα έργα ιδίως του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Υπάρχει και μια άλλη απειλή παντού στην Ευρώπη. Για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζει υψηλό κόστος για να μεταβεί στην ψηφιακή τεχνολογία για να λειτουργήσει στις νέες αυτές αγαρές. Οι ιδιοκτήτες τέτοιων αιθουσών ψάχνουν αξιόλογα έργα κοινή αποδοχής και αυτές οι αίθουσες άμα δεν τύχουν στήριξης, οικονομικής στήριξης τέτοιες αίθουσες που είναι σαν πολιτιστικά κέντρα αντιμετωπίζουν και αυτά πρόβλημα στην αγορά και μπορούν να χαθούν πολύ γρήγορα, να κλείσουν. Θα ήθελα να συστήσω λοιπόν την έκθεση αυτή να την δεχτείτε γιατί είναι μια έκκληση προς όλους, προς τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αρχές, τοπικές και περιφερειακές αρχές προς όλους τους υπεύθυνους για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο ώστε να αντιδράσουν και να δράσουν με συνδυασμένο τρόπο και πιο γρήγορα. Πρέπει να επιταχύνουμε την αντίδραση μας σήμερα για την οικονομική ενίσχυση του κινηματογράφου, ιδιαίτερα για τη μετάβαση του προς τα ψηφιακά. Εμένα δεν φοβίζει το περιεχόμενο γιατί υπάρχει περιεχόμενο ήδη από σήμερα υπάρχει οι διανομής επίσης πρέπει να τύχουν τη στήριξή μας γιατί και αυτοί πρέπει να βρουν τη θέση τους στον ψηφιακό αυτό κόσμο και οι ιδιοκτήτες των αιθουσών δημόσιοι και ιδιώτες Ε, είναι σε θέση που διαφέρει από χώρα σε χώρα και αυτό προτείναμε στην πρότασή μας γιατί διαφορετικά χρηματοδοτικά πρότυπα τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 14 με 20 θα σας δώσω δύο παραδείγματα πρώτον 10 κινηματογράφοι στην Μαλπόλσκα για Κράκοφ και στο Βρότσουαβ στην Πολωνία ως παράδειγμα να δούμε τι έγινε εκεί η μετάβαση σε αυτές τις μικρές πόλεις λόγω των διαρθρωτικών ταμείων μετάβαση προς την ψηφιακή τεχνολογία επέτρεψε στις αίθουσες αυτές να αυξήσουν το κοινό τους κατά 100% και γιατί αυτό διότι τα σινεμά αυτά που ήταν τεράστια μπορούσαν συνήθως έδειχναν αμερικάνικα έργα για μαζικό κοινό μαζί με άλλα ευρωπαϊκά έργα αλλά ταυτόχρονα μπόρεσαν να συνεχίσουν το καθήκον τους στην αποστολή τους να προβάλλουν ευρωπαϊκά έργα κατά 30-40% και έτσι δόθηκε και μεγάλη ευκαιρία επενδύσεων σε αυτές τις μικρές πόλεις. Άλλο σύστημα δεύτερο που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι το λεγόμενο εμπορικό σύστημα για την από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία έκανε μια προτιμησιακή προσφορά για τα ιδιωτικούς κινηματογράφους που επέτρεπε χρηματοδότηση της μετάβασης προς την ψηφιακή τεχνολογία. 80 με 100.000 ευρώ χρειάζονται ανά αίθουσα. Τόσα πίστοση δόθηκε και μέσα σε ένα-δύο χρόνια μπορούσαν οι κινηματογράφοι αίθουσες δηλαδή να το αποπληρώσουν. Αλλιώς θα έκλειναν. Υπάρχει κι άλλο σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει επίσης να γίνει γνωστό και δεν θα το αναφέρω. Άλλο θέμα είναι ένας, υποστηρικτικ... ένας στηρικτικός μηχανισμός συνεννόησης των ιδιοκτητών αιθουσών και καναλιών είναι σύστημα που λειτουργήσε πολύ καλά στις Ηνωμένε Πολιτείε, το VPF. Virtual Print. Καλό σύστημα είναι, καλό. Που επιτρέπει την περικοπή του κόστους της μετάβασης προς την ψηφιακή τεχνολογία. Άλλο θέμα που θέλουμε να θίξουμε στην έκθεση είναι τα πρότυπα. Οι περισσότεροι παραγωγοί και διανομής λένε και ζητάνε από την Κομισιόν νομοθεσία για πρότυπα. Αυτό γίνεται αν υπάρχει ένα εναρμονισμένο σύστημα με τα πρότυπα ίσο. Αλλιώς δημιουργούνται νέοι φραγμοί για τους παραγωγούς διανομής και ιδιοκτήτες αιθουσών. Ενώ αν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα, ένα σύστημα, όπως στις ΗΠΑ και σε μερικές χώρες της Ευρώπης, τότε σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να περικόψουμε, να αφαιρέσουμε τους φραγμούς αυτούς. Ο Ευρωπαίος θεατής το ευρωπαϊκό κοινό ζητάει σήμερα, ζητάει τα συστήματα αυτά 2K ή 4K που επιτρέπουν την προβολή τρισδιάστατων έργων ο Βιμ Βέντερς το έργο του Πίνα το έκανε τρισδιάστατο και αυτό δείχνει πόσο, απαιτητικά είναι, πόσο απαιτητικό είναι σήμερα το κοινό. Η νέα τεχνολογία αφορά τους πάντες παραγωγούς, διανομής και ιδιοκτήτες και πρέπει να υπάρξει τυποποίηση όσο δυνατόν γρηγορότερα γιατί αυτό θα διευκολύνει πολύ τους ιδιοκτήτες των αιθουσών. Υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες που δεν θα τις αναφέρω εδώ σε λεπτομέρεια αλλά τις μάθαμε μέσα, μέσω πολλών συναντήσεών μας με αυτούς. Άλλο πρόβλημα είναι τα αρχεία. Και εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε μία και μόνη απάντηση. Το, τα 35 χιλιοστά κάτω από ορισμένες συνθήκες, τεχνικές, περιβαλλοντικές και το καθεξής αντέχουν ε, πολύ περισσότερο ε, στην ε, ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει τις προδιαγραφές εκείνες που θα μας επιτρέψουν να αρχιοθετήσουμε για πολλά χρόνια τα κινηματογραφικά εκείνα έργα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ε, διδασκαλίας, ε, προαγωγής ε, της έρευνας και το καθεξής. Έτσι λοιπόν η ψηφιοποίηση αυτών των έργων που αυτή τη στιγμή ε, βασίζονται στο αναλογικό σύστημα. Η έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντική αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε την κινηματογραφική μας εκλονομιά για τις μελλοντικές γενιές. Εκ μέρους ε, των κρατών μελών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε την υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν ως ε, στόχο ε, την δημιουργία ταινιωθικών, φιλμωθικών όπως και αν τις ονομάσουμε. Και αυτά ε, είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, ε, κινηματογραφική μας κληρονομιά. Είναι λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, έρχομαι στο ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει η ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο που αντιμετωπίζουμε, που εξετάζουμε στην έκθεση ε, ένα στοιχείο που ανέφεραν και οι Βιμ Μπέντες και οι Ρόμαν Γκούτερκ με τους οποίους ε, συναντήθηκα πριν ε, παρουσιάσω αυτή την έκθεση τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί πρέπει να σας πω ότι πήγα και στο Παρίσι και στο Φεστιβάλ των Κανών. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή πρέπει να αποδώσει σημασία στην ε, κινηματογραφική παιδεία. Για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του Βιμ Βέντες, οι μελλοντικέ γενιές δεν θα πρέπει να είναι ε, εκτεθειμένες ε, σε χειραγωγίες, σε απλουστευτικές παραγωγές. Αναφέρθηκε παλαιότερα από ένα ε, γνωστό κινηματογραφιστή ότι μέσα από τον κινηματογράφο μπορεί κανείς να επηρεάσει ε, τη γλώσσα, ε, τις αρχές. Άρα δηλαδή η κινηματογραφική παιδεία σε επίπεδο κρατών μελών γιατί τα κρατημέλη είναι αρμόδια για τους νέους, αυτή η κινηματογραφική παιδεία πρέπει να ενισχυθεί, να στηριχθεί μέσα από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση. Αυτό βέβαια από την άλλη απαιτεί να υπάρξει και μια μακρόπνοη επένδυση. Αυτό λοιπόν το σύστημα που ε, είναι, βασίζεται σε μια φιλόδοξη κατάσταση ε, λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο σε μια χώρα, στη Γαλλία. Ας έρθουμε τώρα στο πρόγραμμα Media για το οποίο μιλήσαμε. Επιθυμούμε να πούμε προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο ότι το πρόγραμμα Media, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια στηρίζει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, όχι μόνο πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του και τη χρηματοδότησή του, αλλά θα πρέπει να είναι και σε θέση να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, δηλαδή την ψηφιοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων εκείνων που εργάζονται στον κινηματογράφο, κυρίως ε, ε, σε όσους ε, να προετοιμάσει εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιοποίηση. Κατόπιν, το πρόγραμμα πρέπει να αναλάβει και νέες λειτουργίες, δηλαδή τη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μετάφραση κυρίως ε, όλων των ψηφιακών έργων. Ε, το κόστος βέβαια είναι τεράστιο και ίσως ε, μπορούμε να σκεφτούμε και τον υποτιτλισμό γιατί ο μεταγλωτισμός είναι πάρα πολύ δαπανηρός. Πάντως πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Και κατόπιν θα ήθελα να πω ότι πρέπει να στηρίξουμε και τα φεστιβάλ κινηματογράφου αυτά τα φεστιβάλ ε, κινηματογράφου πρέπει να στηριχθούν από όλα τα κρατημέλη. Αυτά θα τα βρείτε όλα ε, στην ε, έκθεσή μου και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μακρηγορήσω περιττέρω από αυτού. Κατόπιν, όσον αφορά το μέλλον των μέσων του κινηματογράφου στην Ευρώπη, Θέλουμε να έχουμε ένα υπεύθυνο μέσο με την έννοια ότι οι υποψήφιοι θεατές να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ε, γραμμικές μεταδόσεις. Επιθυμούμε να φτάσουμε σε έναν ευρωπαϊκό κινηματογράφο ε, που θα έχει όλο και πιο ευρύ ρεπερτόριο και που θα είναι σε θέση να προσελκύει όλο και περισσότερους θεατές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτό το παραδοσιακό σύστημα το οποίο ε, καθίσατε ακόμα πιο σημαντικό με την άφηξη της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Συμφωνώ λοιπόν στο να διατηρήσουμε το γραμμικό σύστημα, αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και σε ένα νέο σύστημα, στο σύστημα των νέων τεχνολογιών. Σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική ε, παραγωγή ε, αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφοι θεατές είναι πάρα πολλοί, αριθμητικά πάρα πολλοί, κατόπιν τούτου πέρα από την υποστήριξη του παραδοσιακού μοντέλου που είναι ε, αιτιολογημένο ε, θα πρέπει να προάγουμε και την εμπορική πτυχή του όλου θέματος που θα επιτρέψει στους θεατές να έχουν μια πολύ πιο ευρεία βεντάλια δυνατοτήτων επιλογής. Επαναλαμβάνω να στηρίξουμε το παραδοσιακό σύστημα και να είμαστε και ανοιχτοί σε καινούργια συστήματα και εδώ βασιζόμαστε στην υποστήριξη των κρατών μελών. Για μας υπάρχει αρκετό περιθώριο και για ε, τα γραμμικά συστήματα αλλά και για εκείνα που είναι πιο κοντά στις ε, νέες τεχνολογίες. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν ε, τις εργασίες που έχουν σχέση με το έργο αυτό, με την εργασία αυτή. Ευχαριστώ όλους ε, όσοι με βοήθησαν. Ε, μπορώ να συναντηθώ βέβαια και με άλλους που ενδιαφέρονται για την έκθεση. Και όσον αφορά την έκθεση αυτή, μπορείτε να βρείτε ίσως και άλλα στοιχεία ε, που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Ε, όμως εκείνο που είναι σημαντικό είναι να εκπέμψουμε ένα χειρό μήνυμα ε, στα κράτη-μέλη και στον κόσμο του κινηματογράφου ότι δηλαδή είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ψηφιακή τεχνολογία που είναι περισσότερο ευκαιρία και λιγότερο πρόκληση ή απειλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς ε, πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε. Τέριαξαν πολύ καλά και με την ε, ακρόαση που έλαβε χώρα. Έχω τώρα δύο παρεμβάσεις, αλλά παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομοι γιατί θα ακολουθήσει αυτή αμέσως οι συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ, αλλά έχουμε κάποιον που διαφέρει τόσο πολύ, είναι τόσο, και κοιτάξε τόσο καλά, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση. 30.000 εργασία ε, φτιάχνει ο Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, μην το υποτιμούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε και πλευρά επιχειρηματική. Είναι ΜΜΕ. Ε, πρέπει να πετύχουν και βασικά το θέμα είναι τι θέλει ο κόσμο, τι ζητάει ο κόσμο. Να μην είμαστε αυθαίρετοι, για το τι, θα, τι ταινίες θα βγαίνουν, αλλά έτσι θα βοηθήσουμε τη γεωματογράφο στην Ευρώπη να προωθούν καλύτερα τις ταινίε και επίσης να ε, αναπτύσσονται κάποιες δεξιότητες, να υπάρχουν το ταλέντο να φτιάχνουμε στην Ευρώπη ε, ταινίε. ακριβώς όπως ε, μας τα είπε ο εισηγητής. Και Και επομένω όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μα για την πολιτική που θα ακολουθεί στο μέλλον. Η πρώτα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η επόμενη. Κοιτάξτε, και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή πολύ υψηλής ποιότητας η έκθεση και νομίζω ότι όσα λέει τα λέει με την καρδιά του τα νιώθει αυτά που γράφει δηλαδή ο εισηγητής όντω θα πρέπει να μπορούμε στο σινεμά να βλέπουμε περισσότερε ευρωπαϊκέ ταινίε και επίση θα πρέπει να ψηφιοποιούνται οι ταινίε και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να ενισχύσουμε τις εξάρτητες παραγωγές ε, αλλά βέβαια για να τα δείξουν κάποιοι μικροί κινηματογράφοι χρειάζονται και αυτή η υποστήριξη. Ε, επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί ο υποτιτλισμός γιατί βοηθά τον κόσμο ε, στη χώρα μου. Φερρυπίν έχουμε ντουμπλάρισμα το οποίο δεν βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης θα ήθελα να σας πω τη γνώμη μου ότι χρειάζεται να βγαίνει κανένα σινεμά γιατί ε, ε, άμα κόσμο πηγαίνει περισσότερο θα έχει περισσότερα χρήματα ο κλάδος και έτσι θα παράγονται περισσότερε ταινίε και θα μπορούμε να καταπονήσουμε και την πειρατεία, ε, τη μαύρη αγορά στο ίντερνετ. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ με αυτή την παροβολή έκθεση θα προωθήσουν τι θέση του Κοινοβουλίου. πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα εντάχει να σας πω πόσο ικανομένη είμαι για αυτή την έκθεση πάρα πολύ εύστοχη, πάρα πολύ καλά φτιαγμένοι, πολύ ενδιαφέρον είναι μαζί να εξετάσουμε τα εξής δύο. Υπήρχε το πρόβλημα της παρέκκλησης εκείνης και λέγαμε ότι το πέρασμα η, πέρασμα, η ενίσχυση στο πέρασμα στην ψηφιακή τεχνολογία θεωρείται κρατική επιδότηση και είχε δοθεί αυτή η παρέκκληση. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε ε, αυτό το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά που αποτελεί αλλαγή πορείας να θεωρηθεί θεμητό το να υπάρχει κρατική στήριξη για αυτές τις αλλαγές όχι μόνο που είναι σημαντικό όπως είπατε τώρα για κινηματογράφους ε, ποιοτικού, αλλά συγκεκριμένη ενίσχυση σε αυτούς που δείχνουν ευρωπαϊκό σινεμά ποιότητας, αλλά επίσης, όπως είπατε, να υπάρχει προσβασιμότητα σε κάποιου είδους πιστώσεις της ε, ΕΤΕ υποτύπων βιομηχανικού δανείου και έτσι να δούμε τις λεπτομέρειες της υποστήριξης για αυτά τα συστήματα όπως το σύστημα το εγκεκριμένο που υπάρχει το ISO, το τυποποιημένο. Αλλά δούμε και το ότι το τρέχον αμερικάνικο σύστημα δεν ταιριάζει, δεν είναι συμβατό με, τις, με τους μικρούς κινηματογράφους. Αυτά επομένω είναι ενδιαφέροντα και πρέπει να μας αποσκοπήσουν Κυρία Τσάιλτερ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μπόρις για την έκθεσή του και αναμένω τη συνεργασία μας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα και για τη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Θα τονίσω ιδιαίτερα μερικές πτυχές όπως τη συνεργασία μεταξύ κινηματογραφιστών, αιθουσών, ολοπικών αρχών και θα ζητήσω χρηματοδότηση των κινηματογραφικών λεσχών. Στη χώρα μου και σε άλλες χώρες οι λέσχες αυτές είναι πολύ μικρού μεγέθους και πρέπει να ενισχυθούν για, τουλάχιστον αρχικά γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία. αλλά φυσικά χρειάζεται να υπάρξει και σαφής ορισμός του τι εννοούμε όταν λέμε εναλλακτικό κινηματογράφος και άλλα. Ο εισηγητής ίσως ξέρει ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο ορισμός, αλλά πρέπει να τον δεχτούμε γενικά. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα χρειάζεται να χειρίζονται τα νέα αυτά μηχανήματα. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν θέλω να προσθέσω ότι η Κομισιόν με το πρόγραμμα ΜΥΔΙΑ πρέπει για το βραβείο Λουξ να φροντίζει και για τον υποτιτλισμό. Πριν από δέκα μέρες είδα στο Βερολίνο και μία βερσιόν ε, κινηματογραφικού έργου για τυφλούς. Μπόρεσαν να πάνε εκεί τυφλοί. Η συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς μου έδειξε ότι είχαν τις ίδιες εντυπώσεις με τους βλέποντες. Πώς γίνεται αφού δεν έβλεπαν. Παρ' όλα αυτά για κάποιον ακατάληπτο λόγο τους άρεσε. Θέλω να πω με αυτό ότι ο υποτιτλισμός είναι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε μία μόνο γλώσσα και όπως είπε και μία ομιλήτρια σε μερικές χώρες υπάρχει πάντα ντουμπλάρισμα σε άλλες μόνο υπότιτλοι. Εμείς είχαμε πάντοτε ντουμπλά στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες πάντοτε υπότιτλους. Το πρόγραμμα Media λοιπόν θα συνεχίσει ελπίζω να χορηγεί περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να αναλάβει και την ιδέα μας και το βραβείο Λούξ να υποτιτλίζεται η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πάκ, δηλαδή κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω αναφερόμενη σε ένα λάθος το μίδια υποστηρίζει και τους υποτίτλους και το ντουμπλάρισμα. Παρόλα αυτά αφήνουμε την επιλογή στον διανομέα και το κατά πόσον θα ζητήσει ντουμπλάρισμα ή υποτίτλους γιατί πιστεύουμε ότι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα για σε ποια αγορά απευθύνονται. Ξέρω ότι το θέμα είναι αμφιλεγόμενο, αλλά υπάρχει και θέμα χρηματοδότησης και διαθεσίμων κοντιλίων μας. Αρχίζω ευχαριστώντας σας για την πρόσκλησή σας, γιατί θέλω να σας πω ότι υποστηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την έκθεση του Πιότρ Μπορίς. Δείχνει τη σημασία που έχει η ψηφιοποίηση ιδιαίτερα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και του τρόπου με τον οποίο η βιομηχανία μας απειλείται αυτή τη στιγμή και πολιορκείται. Η μετάβαση στο ψηφιακό δεν τη χειριζόμαστε όπως έγινε στην τηλεόραση. Περνάμε στο ψηφιακό κινηματογράφο με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα, τα νέα πρότυπα και οι αργές αλλαγές. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά σχόλια που ελπίζω να σας βοηθάνε. Για τα νέα πρότυπα χρηματοδότησης, δυστυχώς, δεν είναι αποδοτικά. Εμείς υποστηρίζουμε την ιδέα του video on demand στα πλαίσια του media. Και μάλιστα Θα έλεγα ότι μερικά από αυτά τα προγράμματα δεν αποσβήνονται παρά μόνο σε τρία χρόνια. Άλλο θέμα. Ό,τι περιτριγυρίζει τις ψηφιακές προβολές. Τον περασμένο Οκτώβριο διαπιστώσαμε ότι παρά το ότι το VPF χρησιμοποιείται ευρέως για τα περισσότερα έργα στην αγορά είναι πιο ακριβό για έναν ευρωπαϊκό διανομέα να διανύμει ψηφιακά ένα έργο από ότι στα 35 χιλιοστά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τη βιομηχανία. <clears throat> Όσο για την ε, εκπαίδευση ως προς το σινεμά. Εμείς στην Κομισιόν δημιουργήσαμε μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τη σύνδεση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ παιδείας και κινηματογραφοφιλίας και καλέσαμε πολλούς ε, εμπειρογνώμονες για να λυθεί αυτό το αδιέξοδο και πράγματι το θέμα των κινηματογραφικών λεσχών παρατηρήθηκε δηλαδή να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα δημιουργίας κινηματογραφικών λεσχών αν το επιτρέψουν τα κονδύλια. Το νέο μίδια θα λύσει ελπίζω ορισμένα από αυτά τα προβλήματα αλλά βλέποντας τις τρέχουσες προτάσεις της Κομισιόν στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα υπάρξουν αρκετά χρήματα για να κάνουμε ούτε τα μισά από όσα είπαμε. Δέχομαι με χαρά την υποστήριξή σας και ελπίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε να έχουμε έναν λογικό τουλάχιστον προϋπολογισμό για τους στόχους μας γιατί ένα από τα κυριότερα προβλήματα για το μέλλον είναι πράγματι η προώθηση του περιεχομένου. Δημιουργούμε πολύ περιεχόμενο και πολλά έργα αλλά υπάρχουν μαζικά έργα και προγράμματα δυστυχώς μόνο οι ισχυρότερες μάρκες, εταιρείες επιλέγονται από τους καταναλωτές και η εμπειρία μας από το DVD που χρειάστηκε να το παρατήσουμε την στηρικτικό μηχανισμό γιατί είχαμε ελπίσει να καταπολεμήσουμε την κυριαρχία της Αμερικής εδώ σημαίνει ότι καταλήξαμε τελικά σε περίπου 25% μερίδιο της αγοράς. Ελπίζουμε στο νέ, στη νέα μορφή VOT και στις νέ, στα νέα επιχειρησιακά πρότυπα να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ αυτού του προγράμματος για να κάνουμε τουλάχιστον μια δοκιμή των νέων αυτών προτύπων. Νομίζουμε όμως ότι τα φεστιβάλ και η διαφήμιση θα είναι το κλειδί. Θα διορθώσω τώρα κάτι. Ο οπτικοακουστικός τομέας απασχολεί 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικός 6 δισεκατομμύρια ευρώ είχε έσοδα πέρυσι και η ετήσια ανάπτυξή του είναι εντυπωσιακή. Τέλος, οι κρατικές επιχορηγήσεις. Φυσικά, συνεχώς κάνουμε διαβούλευση ακόμα με τους ενδιαφέροντες που θα λήξει το Σεπτέμβριο και θα θίξει όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσατε και εσείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Χαιρόμαστε όλος ιδιαιτέρως για τη συνεργασία μας αυτή και πιστεύουμε ότι η έκθεση θα είναι πολύ χρήσιμη για τη σύσταση που ετοιμάζουμε για του χρόνου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, αν θέλει να προσθέσει τίποτα ο εισηγητής, να προσθέσει. Σας ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε. Όλους όσους λάβετε το λόγο σας ευχαριστώ. Όλα αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά θα τα λάβω υπόψη που είπατε. Και πρέπει να σας πω ότι όντως έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το πρόγραμμα αυτό, τα media, το media. Νομίζω ότι είναι καλό το timing, σωστή ώρα ήρθε, διότι α, μετά από το να βλέπει κανείς ταινίες στο σινεμά, το επόμενο βήμα είναι το βίντεο on demand. Σήμερα ακόμα δεν υπάρχει αυτό, και σύμφωνα με όσο είπε η κυρία Πρόεδρος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αναπήρων. Όντως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όντως και αυτό να το εντάξει στην έκθεση. Επίσης, συμφωνώ 100% με την κυρία Κώστα, ότι δηλαδή αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τους κινηματογράφους, τότε χρειάζονται ρυθμίσεις ούτως ώστε να υπάρχει κρατική ενίσχυση. Γιατί λέμε ότι έχουν σημασία κινηματογράφοι και χρηματοδοτούμε τις όπερθες αλλά όχι τον κινηματογράφο. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει όσον αφορά αυτή την κρατική ενίσχυση. Αλλιώς έχουν πρόβλημα κινηματογράφοι, επομένως. Σας τονίζω ότι στον κεις μέλλον για δύο-τρία χρόνια θα πρέπει να έχουμε διτό σύστημα για τους κινηματογράφους. Θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανήματα προβολής ε, παλιωμοδίτικα, αναλογικά, αλλά και ψηφιακά, αν θέλει κανείς να παίξει μια ταινία που έχει γυριστεί πριν από 10-15 χρόνια, ε, ε, δεν θα έχει ψηφιοποιηθεί. Επομένως, σε κάποια σημεία θα πρέπει να έχουμε το διπλό σύστημα. Βέβαια, στο μέλλον Όλα θα είναι ψηφιακά. Όλα. Σας ευχαριστώ για όσα προτείνατε και για όσα είπατε και επομένως ελπίζω ότι όλοι οι μπλεκόμενοι θα λάβουν την ε, γνώμη μας, τη θέση μας και θα αναλάβουν δράση. Το Σεπτέμβριο θα ε, λήξη προθεσμία, έχετε χρόνο για να μπορέσετε να σκεφτείτε, ε, θα έχετε με την ησυχία σας το χρόνο να σκεφτείτε στην παραλία, στο σινεμά, το καλοκαίρι και θα ψηφίσουμε 5 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, επί του παρόντος συμφωνούμε όχι σε όλα, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα θα τη λήξη της συνεδρίασης και σας ευχαριστώ.